Okay, colleagues, good, good afternoon and uh, welcome. Καλημέρα συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα και σημαντικά πράγματα. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να προσθέσω ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη για την επίσκεψη στη Νέα Υόρκη της Επιτροπή μας. Ο τι είναι ο από πλευράς μας του ΕΛΚ. Και αυτό είναι το τελευταίο θέμα για σήμερα. Η ψηφοφορία για την γνωμοδότηση για την κατάσταση στη Μεσόγειο τα θέματα της μετανάστευσης δεν θα γίνει αύριο, αλλά σε μια επόμενη συνεδρίαση στις 10 Νοεμβρίου μάλλον έτσι ώστε να υπάρξει χρόνος για να υπάρξουν συμβιβαστικές γιατί η ΛΥΜΠΕ άλλαξε το χρονοδιαγραμμά της και έτσι έχουμε περισσότερο χρόνο, υπάρχουν σχεδόν 100 τροπολογίες ε, και θα πρέπει να ξεκαθαριστούν καλύτερα τα πράγματα και το μήνυμά μας να είναι και αυτό ξεκάθαρο. Το τελευταίο θέμα σήμερα είναι μια κοινή συνάντηση με το περιβάλλον και τη γεωργία στην 3 σε 50 ή μάλλον έχω κάνει λάθος λέει η πρόεδρος αυτή η συνεδρίαση θα γίνει αύριο όχι σήμερα αύριο είναι μερική διάταξη Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε τελειώσει όλα τα άλλα θέματα πριν πάμε στην συνεδρίαση αύριο το απόγευμα, αυτή την κοινή με τη Λίμπε κτλ. Και επίσης και το θέμα των ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν από τη συνεδρίαση μαζί με την ΕΝΒΗ και την Άγκρη. Λοιπόν, αυτές είναι οι αλλαγές, τις συμφωνείτε. Ευχαριστώ. Κάποιες ανακοινώσεις την 5η, 15 του μηνός, κοινή συνάντηση με την ΑΦΕΤ για την παρουσίαση των υποψηφιωτήτων Βαβίου Σαχάροφ. 9 με 10 και μισή ψηφοφορία για τις υποψηφιότητες και την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, έκτακτη συνεδρίαση, συνάντηση με τον Επίτροπο Μιμίτσα, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τη συνέχεια που θα δοθεί στη Συμφωνία Κοτονού. Θα τα έχει υιοθετήσει τα, τις προτάσεις της μέχρι τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μας τις καταθέσει. Θα σας ενημερώσουμε, εν πάση περιπτώσει, για τις συνεδριάσεις αυτές τις επόμενες μέρες, για να τις λάβετε υπόψη. Λοιπόν, στο τρίτο σημείο είναι έγκριση των πρακτικών. 3η Σεπτεμβρίου, αν έχετε παρατηρήσεις πριν το τέλος συνεδρίασης. Αν δεν πάρουμε προτάσεις αλλαγής θα θεωρηθούν δεκτά τα πρακτικά. Στο 4 τώρα θα βρείτε στο φάκελό σας πάντα τις αποφάσεις και τις συστάσεις των συντονιστών της 22ης Σεπτεμβρίου. Εάν έχετε πάλι κάποιες παρατηρήσεις στη γραμματεία μέχρι το τέλος. Αν δεν πάρουμε παρατηρήσεις τα πρακτικά αυτά θα θεωρηθούν δεκτά. Περνάμε στο 5. Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ένα νέο συνάδελφο, νέο εδώ, τον κύριο Γκριμό. Ο Βενσάν Γκριμό είναι ο νέος σύνδεσμος ανάμεσα στην Επιτροπή και την ε, δική μας Επιτροπή. Και έχει και μία συνάδελφό του μαζί, την κυρία Παύλικ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή που κάνατε. Είμαι υπεύθυνο για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο στη Γενική Διεύθυνση και με χαρά θα συνδιαλαγώ μαζί σας. Την προηγούμενη εβδομάδα υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόταση για την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης official step in this uh, process and it is meant uh, not to take και τον χρόνο SCB. Προς το παρόν δεν ε, προτείνουμε να καταλήξουμε σε μια θέση αλλά θέλουμε να ξεκινήσουμε ε, μια διαβούλευση για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων ε, με δεκτικό τρόπο. Ο κύριος Μίμητσα θα σας τα παρουσιάσει όλα αυτά με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες τη Δευτέρα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Πολύ σημαντική συνάντηση αυτή. Την Δευτέρα θα μας τα πει ο Επίτροπος. Και καλώς ορίσατε κύριε Γκριμό. Περνάω λοιπόν στο 6 θέματα εκπαίδευσης των παιδιών σε καταστάσεις ε, κατεπίγουσες. Ε, ξέρετε ότι πριν από το καλοκαίρι αποφασίσαμε να προετοιμάσουμε μια προφορική ερώτηση με ψήφισμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπαίδευση των παιδιών σε κατεπίγουσες καταστάσεις. Θα ψηφίσουμε για την έκθεση αυτή στη συνάντησή μας της 10 Νοεμβρίου Νομίζω ότι το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει, τα προβλήματα δηλαδή που αντιμετωπίζουν τα παιδιά πρόσφυγες. Και θα τεθεί αυτό το θέμα και μετά την επίσκεψη στην Τουρκία που θα συζητήσουμε αμέσως μετά. Τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και η έλλειψη εκπαίδευσης. Έχω στην εκλογική μου περιφέρεια κάποιον ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει κανένα από τα στάδια της εκπαίδευσης ακριβώς γιατί είναι πρόσφυγας από την Σομαλία και είναι 20 ετών. Και ένα από τα προβλήματα και ένας από τους λόγους για τους οποίους εγκαταλείπουν τις χώρες τους οι άνθρωποι αυτοί και τη Συρία είναι ακριβώς η έλλειψη εκπαίδευσης και σε αυτές τις χώρες και σε αυτή τη χώρα και αναφέρομαι εδώ στα παιδιά τα οποία σπουδάζουν και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Λοιπόν ζητάμε σε επίπεδο δημοσιονομικό να αυξηθεί η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση των παιδιών. Ξέρω ότι ο Επίτροπος Τηλιανίδης μας έχει πει ότι θα υποστηρίξει τις προτινόμενες αλλαγές και εμείς στα πλαίσια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό θέλουμε να υπάρξει μια κάποια αύξηση και να υπάρξει μια θετική αλλαγή. Είναι χρήσιμο όμως σε αυτό το πλαίσιο να γίνει μια συζήτηση σήμερα με εμπειρογνώμονες και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από ΜΚΟ και από τα Ηνωμένα Έθνη που εμπλέκονται σε θέματα εκπαίδευσης, εκπαίδευσης παιδιών σε κατεπίγουσες καταστάσεις. Σκίνερ, διευθύντρια της ε, UNICEF, Λέτζου από την ΕΚΟ, υπεύθυνη για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την θέση των παιδιών στις συγκρούσεις, διεθνείς συγκρούσεις. Λορέντσο, Δεύκο. Και έχουμε επίσης και από τη ΜΚΟ World Vision εκπρόσωπο. Δέκα λεπτά η καθεμία και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση με τους συναδέλφους. Η κυρία Σκίνερ από τη UNICEF. Εμείς πήγαμε στην Τουρκία και είδαμε την εξαιρετική δουλειά την οποία κάνει η UNICEF στα στρατόπεδα και στους καταβλισμούς εκεί. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους σας συναδελφοί. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ. Είμαι καινούργια εδώ στις Βρυξέλλες ως ε, διευθυντρία της UNICEF σε σχέση με τις, ε, τα θεσμικά όργανα και θα πρέπει να σας πω ότι έχω ε, δουλέψει και στο Μαυροβούνιο, αλλά πάντα αυτό που με απασχολούσε πιο πολύ στην καριέρα μου στη UNICEF ήταν η εκπαίδευση. Στην πρώτη μου θέση πριν από 15 χρόνια ως υπεύθυνη για θέματα εκπαίδευση στο Κωσυφοπέδιο μετά τον πόλεμο συνεργαστήκαμε με τις αρχές για να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα, ένα σύστημα παιδείας, εκπαίδευσης μετά τον πόλεμο. Επίσης, ε, με στείλαν στην ΑΕΤ μετά τον σεισμό για να υποστηρίξω την ε, όλη προσπάθεια που έγινε για τα θέματα εκπαίδευσης και πρέπει να σας πω από πρώτο χέρι ότι πρόκειται για μια παρέμβαση που σώζει ζωές. Η παροχή δηλαδή η εκπαίδευση σε τέτοιε καταστάσει έκτακτη ανάγκη μετά από συγκρούσει, μετά από πολέμου, μετά από φυσικέ καταστροφέ. Πραγματικά υπάρχει μια διάσταση που σώζει ζωέ. Δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Με απασχολεί λοιπόν πάρα πολύ το θέμα αυτό και χαίρομαι που ε, παίρνω το λόγο ενώπιον τη Επιτροπή σα γι' αυτό. Κάποια αρνητικά στοιχεία επιτρέψτε μου όταν κοιτάμε συνολικά. Όλα τα παιδιά τα οποία είναι σε ηλικία δημοτικού. 6 έως 11 βλέπουμε 5 εκατομμύρια, 50 ε, εκατομμύρια παιδιά τα οποία δεν πάνε στο σχολείο, στο δημοτικό. Και 60 ε, εκατομμύρια ε, εφήβους που δεν πηγαίνουν στο σχολείο. 43% όλων των παιδιών που δεν πηγαίνουν στο σχολείο είναι από χώρες όπου, ε, που έχουν πληχθεί από ανθρωπιστικές κρίσεις. Ε, οι γυναίκες είναι ε, κατά 90% πιο πιθανόν να μην παρακολουθήσουν το γυμνάσιο και λυκείο σε σχέση με τα γόρια. Στη Μέση Ανατολή 46 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε κατάσταση εξαιρετικού ανάγκης. 28,6 εκατομμύρια σε ηλικία 6 έως 11 και 15 εκατομμύρια παιδιά στη Μέση Ανατολή δεν πάνε στο σχολείο. Πραγματικά ε, η εκπαίδευση υποτιμάται. 2,7 εκατομμύρια στη Συρία δεν πηγαίνουν στο σχολείο, 6% στην Ιεμένη. Αντίστοιχα τα ποσοστά και στη Σουδάν. Και μπορώ να συνεχίσω χωρίς τέλος. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα αριθμητικά στοιχεία. Κινδυνεύουμε να χάσουμε μια ολόκληρη γενιά μεταξύ των ε, κρίσεων και των συγκρούσεων που πλήττουν Υπάρχει λοιπόν ε, μεγάλη ανάγκη για αλληλεγγύη στα παιδιά αυτά. Και όπως σας είπα, ε, πρόκειται για μια δραστηριότητα που σώσει ζωές. Ε, η εκπαίδευση μπορεί να προστατεύσει σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Μπορεί να δώσει μια αίσθηση κανονικότητας ακόμα και στις πλέον εξαιρετικές καταστάσεις. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και καινοτόμε τακτικές. Ένα σχολείο μπορεί επίσης να δώσει και άλλα πράγματα όπως ε, φαγητό, ε, υγειονομική περίθαλψη, κάποια βασική, κάποιες βασικές ικανότητες, ε, κάποια ενίσχυση της αντοχής και της ανθεκτικότητας των νέων. Και το συνολικό, η συνολική χρηματοδότηση για την εκπαίδευση έχει μειωθεί. Έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση για την εκπαίδευση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκες. 39 δις ευρώ δολάρια. Τα χρειάζονταν όμως, έχουμε υπολογίσει, για να πετύχει το STD4, ο ρωσοκόσμος, δηλαδή ένα ε, ίσο επίπεδο εκπαίδευσης. Και αυτό περιλαμβάνει και τις καταστάσεις εκτάξεων ανάγκης και παρατεταμένης κρίσης. Για να φτάσουμε δηλαδή σε ένα επίπεδο ανθρωπιστικό αποδεκτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αναγνωρίζει τη σημασία τη ε, χρηματοδότησης τη εκπαίδευση σε κατάσταση καταστάσεις και καλωσορίζουμε την πρόταση αύξηση ε, των ε, ποσών χρηματοδότηση αυτής. Καλωσορίζουμε επίσης τη δημιουργία καταπιστευμάτων και επίσης σημειώνουμε ότι μία πρώτη τέτοια παρέμβαση ήταν αυτή τη UNICEF στην Τουρκία και αναφέρατε και εσεί πρόεδρε τι γίνεται επί τόπου. Καλωσορίζουμε επίση την έκκληση και την όθηση από την Επιτροπή σα για την αύξηση πόρων και χρηματοδότηση σε εκπαίδευση σε εκτακτή, σε σε καταστάσει. Η UNICEF αποτελεί μία οργάνωση η οποία έχει μεγάλη εμπειρία. Βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά της κρίσης. Ε, γίνεται μια σωστή αξιολόγηση με ε, τυπικό και μη τυπικό τρόπο. Η, τα παιδιά είναι τα πιο ευάλωτα άτομα σε τέτοιες καταστάσεις. Η επένδυση λοιπόν στην εκπαίδευση σημαίνει εκπαίδευση επένδυση στα παιδιά, επένδυση στην ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει Πέτρος, και σας ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρονικό όριο για να μας δείξετε την κλίμακα του προβλήματος που είναι πραγματικά τεράστια. Είναι πραγματικά πολύ πολύ τα πράγματα και στην Τουρκία. Ένα θέμα ήταν, για παράδειγμα, το κατά πόσο τα παιδιά στην Συρία θα έπρεπε να ακολουθήσουν το σχολικό πρόγραμμα της Συρίας. Ήταν πραγματικό θέμα αυτό. Ή θα έπρεπε μήπω να ακολουθήσουν το τουρκικό πρόγραμμα, μια και θα μένουν πολλά χρόνια στην Τουρκία. Υπάρχουν λοιπόν πολύ σύνθετα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν και θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε πώ επιλύονται. Επόμενη ομιλήτρια. Η Μαρία Λέτζου από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Υπεύθυνη για την προστασία των παιδιών σε ένοπλες σειράξεις και έχουμε επισημάνει το θέμα της χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανακύπτει κάθε φορά που συνομιλούμε με κάποιους φορείς. Η ανθρωπιστική βοήθεια δίνει ενδεχομένως τη μακροπρόθεμη διάσταση που χρειάζονται στην ΕΦΚΟ. Ελπίζω να μας καθησυχάσετε ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία. Να ακούσουμε λοιπόν ποια θα είναι τα αποτελέσματα και πώς μπορούν να επιληθούν τα τεχνικά προβλήματα. Η κυρία Λέβη λοιπόν έχει το λόγο. Thank you very Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ που μας ε, δίνετε τη δυνατότητα για να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα ε, σήμερα. Και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τις ερωτήσεις μαζί με τους ε, συναδέλφους. Παρακαλώ πρώτη διαφάνεια. Παρά το γεγονός ότι η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες δικαίωμα για όλα τα παιδιά, πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ένα 2% του προϋπολογισμού, του παγκόσμιου προϋπολογισμού πηγαίνει στην εκπαίδευση, ίσως και λίγο λιγότερο από το 2% ενώ η εκπαίδευση είναι ύψης της σημασίας για το μέλλον των παιδιών. Με την κρίση της μετανάστευσης πολλά παιδιά ε, φεύγουν όχι μόνο για να έχουν ε, φαγητό και τροφή γενικά, αλλά και το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η UNICEF ε, μας εξήγησε πολύ καλά γιατί έχει σημασία η εκπαίδευση, δεν θα επεκταθώ. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, ε, χάρη ε, στο, στο βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη που δόθηκε στα Ηνωμένα Έθνη του 2012, προωθεί την ε, πρωτοβουλία ειρήνης για τα παιδιά. Από το 2012 αυτή η πρωτοβουλία αυξάνεται κάθε χρόνο και έχουμε δώσει 23 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, άρα θα φτάσουμε στα 1,5 εκατομμύρια παιδιά σε όλες τις ε, χώρες ανά τον κόσμο. Το 2015 ε, έχουμε εγγράψει 20 εκατομμύρια σε 16 projects και προσθέσαμε και 1 εκατομμύριο για τα παιδιά που είχαν πληγεί από τον ιό έμπολα και δεν είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση εξαιτία της επιδημίας αυτή. Αυτό το πρόθεσε η UNICEF μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Save the Children. Επειδή η κρίση ολοένα και παρατείνεται, θα πρέπει να υποστηρίξουμε πολύ περισσότερο την εκπαίδευση. Γι' αυτό ο Επίτροπος Τηλιανίδης ανακοίνωσε την πρόθεση του να κλιμακώσει τη βοήθεια προς την εκπαίδευση έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα 4% του ανθρωπιστικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια της θητείας. Έχει ξεκινήσει συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη για αυτή την επιπρόσθετη χρηματοδότηση και οι σοσιαλιστές και δημοκράτες και άλλες ε, ομάδες ζήτησαν 26 εκατομμύρια επιπροσθέτως, ε, δηλαδή για το 2016. Παρόλα αυτά, η εκπαίδευση αφορά όλους. Έχουν ευθύνη για αυτήν όλοι οι φορείς γιατί πρόκειται για ένα μακροχρόνιο, για μια μακροχρόνια προοπτική. Γι' αυτό η χρηματοδότηση αναπτυξιακού χαρακτήρα θα πρέπει να προωθηθεί στον τομέα της εκπαίδευσης. Η συνάδελφος από την ΤΕΒΚΟ θα σας δώσει λεπτομέρειες. Ήδη εργαζόμαστε με τους συναδέλφους από την ΤΕΒΚΟ έτσι ώστε να υπάρξει ε, ένα πρόγραμμα σύνθετης χρηματοδότησης και αυτό το συζητήσαμε μέσα στα πλαίσια των ε, καταστάσεων επίγουσας ανάγκης. Και επίσης έγινε ε, μία κοινή σύμπραξη ΕΚΟ και που συνόδευσε τον κύριο Στυλιανίδη το απόγευμα, το καλοκαίρι με συγχωρείτε, στο Ελσίνκι. Επίσης υπήρξε συνεχής χρηματοδότηση από τα μέσα χρηματοδότησης, δηλαδή η UNICEF στην Τουρκία, για παράδειγμα, δέχτηκε χρηματοδότηση του, το 2014 έτσι ώστε να υπάρχει εκπαίδευση για τους ε, Σύριους πρόσφυγες στους καταβλισμούς. Επίσης, στο Μιανμάρ υπάρχει ένα πρόγραμμα μέσα στα πλαίσια του 13 όπου συνέπραξε και η Εκκλησία για να βοηθήσουμε ε, τα παιδιά στο Μιανμάρ και στο Ραγκούν μέσα στα πλαίσια και της κατάρτισης των δασκάλων. Παράλληλα μιλήσαμε για 2.000 εκατομμύρια μεταξύ 15 και 17. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς αυτό το πρόγραμμα επιτυχίας μπορεί να δημιουργήσει διασυνδέσεις και η ΤΕΦΚΟ και ΕΚΟ συνεργάζονται έτσι ώστε στο ετήσιο σεμινάριο της ΔΕΦΚΟ θα συζητήσει εστιακά σημεία σε σχέση με αυτούς τους συνδέσμους που πρέπει να δημιουργηθούν. Σας ευχαριστώ. Ε, Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ, κυρία Λορέντσο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα που αφορά τον ε, ρόλο της συνεργασίας στην εκπαίδευση. Ίσως ο τίτλος του ψηφίσματος δεν θα πρέπει να αφορά την εκπαίδευση σε καταστάσεις επίγουσας ανάγκης, αλλά να μιλάμε για ε, παρατεταμένη κρίση γιατί αυτές, αυτές οι επίγουσες ανάγκες, η επίγουσα κατάσταση αποκτά χρόνιο χαρακτήρα. Και πολλές φορές προσφέρουμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε καταβλισμούς για 10, 15 και 20 χρόνια. Γι' αυτό θα πρέπει να συνδράμει η ανάπτυξη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού για ανθρωπιστικές ανάγκες ένα από τα πιο βασικά ζητήματα είναι πώς να μειωθεί ε, αυτό, αυτός ο φραγμός, αυτό το φράγμα που υπάρχει μεταξύ ανάπτυξης και προανθρωπιστικών προγραμμάτων, διότι μιλάμε για πρόσφυγες που έχουν τις ίδιες ε, ανάγκες, ζουν υπό παρόμοιες συνθήκες και έμπρακτα αυτό που αντιμετωπίσουμε σήμερα σαν πρόβλημα είναι πώς να διαρθρώσουμε τα διάφορα μέσα έτσι ε, ώστε να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση και να μην κάνουμε και κακό. Έχω ορισμένες διαφάνειες να σας δείξω. Για να δείτε τι κάνουμε στον τομέα της εκπαίδευσης ιδιαίτερα για τα ευάλωτα κράτη, για να σας δώσω και μία τάξη μεγέθους, για να δείτε πώς έχουν ή πώς διαμορφώνται οι επενδύσεις μέσα στα πλαίσια του πολιετούς και να μιλήσουμε και για μηχανισμούς στη συνέχεια, γιατί μας απασχολούν ιδιαίτερα. Στο αναπτυξιακό δίκτυο. Το 2014-2015 η υποστήριξη της εκπαίδευσης είναι ε, πολύ σημαντική και εάν δείτε στην επόμενη διαπάνεια βλέπετε ότι συνολικά υπάρχει ανωδική τάση σε σχέση με το προηγούμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. και παρά το γεγονός ότι η, ανώτατη, η ανώτερη εκπαίδευση δεν λαμβάνεται υπόψη, αυτό που έχει σημασία ε, είναι τα περιφερειακά προγράμματα και οι θεματικές γραμμές. Στη συνέχεια βλέπετε την γεωγραφική κατανομή. Έχουμε 39 χώρες ε, όπου εστιάζουμε την προσοχή μας και το 15% το ίμιση e δηλαδή ε, που είναι υπογραμμισμένες με κόκκινο είναι ευάλωτες χώρες. Μιλάμε για 2,7 δις και το 60% προορίζεται για τις ε, ευάλωτες χώρες. Υπάρχουν και διάφοροι υποτομείς Άρα μιλάμε για τη βασική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Επίσης υπάρχει επιμερισμός, η κατανομή μεταξύ Αφρικής και Ασίας. Το 85% στοχεύει τα διμερή προγράμματα και το 15% αφορά την ε, παγκόσμια εταιρική σχέση για την εκπαίδευση. Μέσα στα πλαίσια της ε, συνολικής αυτής ε, εταιρικής σχέσης, παγκόσμιας εταιρικής σχέσης, ε, υπάρχει κατανομή ιδιαίτερα προς τις ευάλωτες χώρες όπου ο προϋπολογισμός έχει αυξηθεί από 21-49%. Αυτό ήταν απόρρια των κρίσεων και της ευαλωτότητας αυτών των κρατών. το GP είχε χρηματοδοτήσει κατά ένα δις ε, δολάρια τις ευάλωτες χώρες. Αν τώρα μιλήσουμε τον, ε, το σημείο διαπαφής ε, μεταξύ των, της κοινή ευθύνης και των παρατεταμένων κρίσεων, βλέπετε ότι η ΔΕΒΟ ασχολείται με την εφαρμογή και τις πρακτικές επιπτώσεις. Θα μιλήσω για τους μηχανισμούς που στην ουσία έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Και αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε ένα προγραμματισμό ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Δεν υπάρχουν συνολικές λύσεις θα πρέπει να εστιάζονται αναχώρα και όταν αποστέλλονται ε, αντιπροσωπείες και στα γραφεία της ΕΚΟ υπάρχει συνεργασία έτσι ώστε να δούμε πόσο ορίζονται οι μηχανισμοί παρέμβασης, άρα οι ΕΚΟ μπορεί να δράσει άμεσα για 12-18 μήνες ανάλογα. Και μπορούμε να αναλάβουμε και τη χρηματοδότηση μετά. Αλλά όλα αυτά βασίζονται σε έναν ad hoc μηχανισμό και σε ορισμένα σημεία της γης. Θα πρέπει όμως ε, να υπάρχουν πιο ε, συστηματικές συμφωνίες μεταξύ ΕΚΟ και ΔΕΒΕ και Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε πολύ καλά παραδείγματα, επιτόπια παραδείγματα, χωρίς να υπάρχει πάντα σωστή τεκμηρίωση. Θα πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες στο περιφερειακό πρόγραμμα της Ασίας. Ε, έχουμε την βοήθεια προς, προς που έχουν ε, μετατοπιστεί ή εκτοπιστεί. Υποστηρίζουμε τα, ε, τους καταβλισμούς στην Ταϊλάνδη τα τελευταία 15-20 χρόνια και τα τελευταία 5 χρόνια εστιάσαμε την προσοχή μας στην εκπαίδευση γιατί αυτό έχει σημασία για την ε, ε, επανεισδοχή αυτής της νέας γενιάς, ε, την επάνωδο στην, στη, στο Μιανμάρ. Ένα άλλο παράδειγμα το βλέπετε στα ε, διάφορα ε, ταμεία ε, καταπίστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν υπάρχει πια αυτό, αυτός ο φραγμός μεταξύ ανθρωπιστικής ε, βοήθειας και Ντεύκο, Βλέπετε το Μπεκού Trust Fund, το, Μαντάντ, το Ταμείο Μαντάντ και το Ταμείο Έκτακτης ε, Ανάγκης για την Αφρική. Μετά μιλάμε για την συνολική εταιρική σχέση για την εκπαίδευση που έχει μεγάλη σημασία σε περίπτωση σύραξης γιατί μπορεί αυτόματα να, να επιδοθεί ένα 20% της τρέχουσας χρηματοδότησης μέσα στα πλαίσια ενδεικτικών πλαισίων. ξεκίνησε στη, στο Νότιο Σουδάν και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Μιλάμε για 30 και 50 εκατομμύρια δολάρια. Το 20% βεβαίως είναι αρκετά περιορισμένο, αλλά ίσως βρούμε και επιπρόσθετους μηχανισμούς. Τέλος, το σχέδιο ψηφίσματος μιλάτε και εσείς για την κοινή πλατφόρμα για την εκπαίδευση όπου θα πρέπει να συμμετέχουμε και εμείς. Εδώ συμμετέχουν πολλαπλοί δωρητές και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα κενά χρηματοδότησης, ποιο είναι το χάσμα μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προσκόμματα ή αυτά τα χάσματα μέσα από μια κοινή πλατφόρμα για να δοθεί μια συνέχεια. Μιλάμε λοιπόν για ένα ανθρωπιστικό ταμείο για την εκπαίδευση. Το βλέπουμε σε επίπεδο τεχνικής ομάδας και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε φτάσει σε μία σαφή πλατφόρμα. Νομίζω ότι θα δοθούν μεγάλες ευκαιρίες από το, από το Global Partnership. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει ανάδραση από αυτή τη μελέτη η οποία χρηματοδοτείται τώρα και θα επιδοθεί στην Κομισιόν. Ε, μιλάτε για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει πληθώρα πρωτοβολιών και θα θέλαμε να ξέρουμε πώς ε, συνδέονται γιατί στη Νέα Υόρκη έγινε λόγος για μία άλλη πρωτοβουλία. Έτσι μας είπαν η Δανή Πρωθυπουργός, ε, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου της Αυστραλίας. Υπάρχουν ε, πολλές πρωτοβουλίες και από τον ιδιωτικό τομέα και δεν ξέρω πώς όλα αυτά εντάσσονται το ένα στο άλλο. Ακούσαμε το θεσμικό πλαίσιο. Πώς το, πώς το είδατε επιτοπίως, πώς εργαστήκατε. Ευχαριστώ. Λέγομαι Λούση. Εκπροσωπώ της ΜΚΟ. Έχω εκπαιδευτεί σε θέματα κατεπηγουσών καταστάσεων και θα μπορέσω να σας μεταφέρω λίγο την εικόνα που ε, επικρατεί επιτόπου στους καταβλισμούς. Έχω περάσει πάρα πολύ χρόνο στην δημιουργία προγραμμάτων εκπαιδευτικών στο βόρειο Ιράκ, στις περιοχές που γειτονεύουν με τις περιοχές που κατέχονται από το ίσις. Νομίζω ότι σωστά αναφερθήκατε στα θέματα προστασίας και στην παράταση γενικά της παραμονής των προσφύγων στους καταβλισμούς αυτούς ο μέσος όρος είναι 17 χρόνια, δηλαδή περίπου η διάρκεια ζωής ε, ενός, ε, η διάρκεια ζωής ε, εννοώ στην παιδική ηλικία ενός ανθρώπου. Οπότε τίθεται το θέμα της εκπαίδευσης και αναφερόμαστε σε ποιοτική εκπαίδευση και προστασία ταυτόχρονα. Γιατί η εκπαίδευση είναι ένα μέσο για την προστασία. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση. Νομίζω ότι έχει σημασία να κατανοήσουμε τις ε, κατεπίγουσες καταστάσεις επίπεδου 3 που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα. Έχουμε χρονίζουσες κρίσεις και καταστροφές τελευταία πρόσφατες. Είχαμε, αν θέλετε, το 2013 τον τυφώνα στις Φιλιππίνες. Ξέρετε τι έγινε στο Νεπάλ που είχα πάει και τον Απρίλιο του προηγούμενου χρόνου. Έχουμε την χρονίζουσα κρίση στην Συρία, στην Τουρκία, Λίβανο, Ιορδανία, Ιράκ. Έχουμε χρόνιες κρίσεις στο Νότιο Σουδάν, όπως επίσης και στον Ήγυρα και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Συνεπώς λοιπόν στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα στην εκπαίδευση ουσιαστικά αγνοείται γιατί δεν έχουμε τα απαιτούμενα χρήματα για να καλύψουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών αυτών των προσφύγων. Τα θέματα της εκπαίδευσης είναι περίπλοκα φυσικά, το δέχομαι αυτό. Υπάρχουν προβλήματα προγράμματος, υπάρχουν προβλήματα γλώσσας, κουλτούρας κτλ. Θα ήθελα εγώ να μιλήσω λίγο τώρα για τα παιδιά, για τη φωνή των παιδιών. Η οργάνωση World Vision έχει εργαστεί πολύ στα πλαίσια προσπαθειών συνολικότερων της UNICEF πρωταγωνιστήσαμε θα έλεγα στην τελευταία συνάντηση ε, των ε, ΜΚΙΟ. Εκπαιδεύσαμε 6.000 παιδιά και τα παιδιά τα ταυτοποιήσαμε και συστηματοποιήσαμε τα θέματα της εκπαίδευσής τους και της προστασία τους και σε τοπικές κρίσεις και σε παρατηνόμενες φυσικά ε, κρίσεις και σειράξεις. Εμείς προσπαθούμε να δούμε τι θέλουν τα παιδιά, δηλαδή τι θέλουν οι κοινότητες. Υπάρχει και η πρωτοβουλία για την ειρήνη και τα παιδιά. Πρόκειται για ένα έγγραφο με συγκεκριμένες διεκδικητικές θέσεις για το Νότιο Σουδάν, την Αιθιοπία και άλλες χώρες. Γενικά ο κοινός μύτος όλων αυτών των περιπτώσεων είναι η σωστή προτεραιότητα και αξιολόγηση του αιτήματο για εκπαίδευση, της ανάγκης για εκπαίδευση. Στη μελέτη για την κεντροαφρικανική δημοκρατία οι γονείς πιστεύουν ότι μαζί με την υγεία, το νερό και την προστασία φυσικά και την κατοικία είναι στο ίδιο επίπεδο. Δεν μπορούμε μόνο με τα τρόφιμα να καλύψουμε τις ανάγκες. Στο σχολείο μαθαίνω, στο σχολείο νιώθω καλά, νιώθω κανονικός, και ε, ακούγονται τα παιδιά, ακούγονται οι κοινότητες και γι' αυτό αυτή τη φωνή ε, πρέπει να την ακούμε και σε τέτοιου είδους φόρα. Τώρα για, για το Βόρειο Ιράκ, ε, η World Vision εκεί έχει μια ολοκληρωμένη προσφορά εκπαιδευτική και σε προσωρινές κοινότητες και σε μόνιμους καταβλισμούς. Έχουμε επίσης και την εκστρατεία Back to School, πίσω στο σχολείο. Πολλές φορές τα παιδιά όταν δεν μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο παντρεύονται πάρα πολύ νωρίς και δεν είναι το μέλλον που επιθυμούν τα κορίτσια κυρίως γι' αυτό. Συνεπώς λοιπόν όταν τα κορίτσια ολοκληρώνουν την εκπαιδευτική τους διαδικασία ε, έχουν πολλά να προσφέρουν στην κοινωνική συνοχή και στην ειρήνη. Δημιουργικά λοιπόν βλέπουμε την εκπαίδευση σαν πολλαπλασιαστή των στόχων ανάπτυξης. Λοιπόν, σε σχέση τώρα με συγκεκριμένα στοιχεία θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να συλλέξουμε περισσότερα στοιχεία για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και να πείσουμε. Υπάρχουν πολλές φαιές περιοχές οι οποίες δεν έχουν τεκμηριωθεί ακόμα. Εγώ βλέπω σε καθημερινή βάση στη δουλειά μου τι ανάγκες υπάρχουν, τι ανάγκες δεν καλύπτουμε και γι' αυτό πρέπει με πολλή προσοχή εμείς να τεκμηριώνουμε το τι κάνουμε γιατί αυτό επηρεάζει θετικά τη ζωή των κοινοτήτων συνολικά. Η κοινότητα των ΜΚΟ λοιπόν καλωσορίζει την προσπάθεια του Επιτρόπου Στυλιανίδη ε, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα την αντιμετώπιση των κατεπηγουσών ε, καταστάσεων. Ε, αυτό είναι το ελάχιστο το 4%. Εμείς θέλουμε ευέλικτα πολυετή συστήματα χρηματοδότησης της εκπαίδευσης. Αυτό είναι ο βασικός στόχος που έχουμε εμείς. χρηματοδότηση για ένα χρόνο δεν φτάνει. Εμείς στο Βόρειο Ιράκ θέλουμε να υπάρξει μια προγραμματική περίοδος χρηματοδότησης. Εμείς δείχνουμε την ανάγκη που έχουν τα παιδιά να, να πάρουν ε, στοιχεία εκπαίδευσης αλλά να συνδεθούν και με μια κάποια προοπτική έτσι ώστε τα παιδιά ε, με τα οποία εργαζόμαστε, με τα ατυπικά προγράμματα, να μπορέσουν να ενταχθούν στο κανονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα έτσι ώστε η εκπαιδευτική τους διαδικασία να επισημοποιηθεί, να επικυρωθεί, να αναγνωριστεί επίσημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σαν δρόντες επιτόπου και δρόσες επιτόπου προσπαθούμε ε, να προωθήσουμε. Εμείς θέλουμε να επικυρώσουν ε, και να εγκρίνουμε με επίσημα χαρτιά την εκπαίδευση που παίρνουν όπως και την εκπαίδευση που παίρνουν οι δάσκαλοι. Έτσι όταν, όταν γυρίσουν στη Σομαλία η εκπαίδευση την οποία παίρνουν να έχουν κάτι να κάνουν με αυτήν. Θα είμαι γρήγορη λέω μιλήτρια. I think we focused a lot on protraction on crisis. Λοιπόν για την παράταση των κρίσεων Έχοντας ε, ξοδέψει αρκετό χρόνο στο Χαγιάν της Φιλιππίνες μετά από τον τυφώνα, ε, είδαμε και επίσης τι συμβαίνει με τους σεισμούς στο Νεπάλ, βλέπουμε πώς λειτουργούν, οι καταστροφές και οι κατεπίγουσες καταστάσεις που δημιουργούνται μετά τη λήξη των πρώτων κατεπίγουσων καταστάσεων. Εμείς λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να προετοιμάζονται σωστά οι κοινότητες, να γίνονται πιο ανεκτές οι κοινότητες, τα προγράμματα λοιπόν αύξησης της αντοχής ε, των τοπικών πληθυσμών σε φυσικές καταστροφές είναι κάτι το οποίο προωθούμε σε κάθε σχολείο και κάθε νέο σχολείο στον Νεπάλ είναι ένα ασφαλές αντισυσμικό σχολείο ε, Ευτυχώς στο Νεπάλ ε, ο σεισμός έγινε στιγμή που δεν ήταν τα παιδιά στο σχολείο. Ε, στην Αϊτή με τον σεισμό ε, δυστυχώς τα κτίρια και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας κατέρευσαν και πολλά σχολεία κατέρευσαν με θλιβερές συνέπειες. Ευτυχώς όμως στο Νεπάλ δεν συνέβη κάτι τέτοιο και η διαδικασία ανάκαμψης είναι μια διαδικασία θα έλεγα καλή. Τώρα, ε, ε, εξόδεψα πολύ χρόνο. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι βλέπω ότι έχει υπάρξει μια συμφωνία έτσι ώστε αυτό το ελάχιστο 4% στην αύξηση των ποσών να γίνει πραγματικότητα. Είναι το ελάχιστο δυνατό. Θα πρέπει ένας μηχανισμός να δημιουργηθεί για σωστότερες σχέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις ΜΚΟ, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν κρατικές υποδομές, σε εύθραστες περιοχές. Συνεργασία και με τα Ηνωμένα Έθνη και με το Νορβηγικό Ταμείο για τους Πρόσφυγες για να βοηθήσουμε την εκπαίδευση σε παρατηνόμενες κρίσεις έτσι ώστε να διασφαλίσουμε χρηματοδότηση προβλέψιμη για ποιοτική εκπαίδευση, για ευκαιρίες μάθησης για τα παιδιά και τη νεότητα γενικά. Και η νεότητα είναι θέμα. Πρόκειται για μια κοινωνική κατηγορία η οποία δυστυχώς δεν μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα μέχρι τώρα και είναι σημαντική και ευαίσθητη. Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης είναι μια επένδυση θα έλεγα, δεν είναι μια δαπάνη. Παρέχει προστασία, σώζει ζωές και επιτρέπει στα παιδιά να μεγαλώσουν, να ανακάμψουν να ανθίσουν ακόμα και στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα και εδώ τίθεται το θέμα <clears throat> της αντοχής, της ανθεκτικότητας, να μπορέσουν να ξεπεράσουν δυσκολίες τα παιδιά. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι τα παιδιά να υποστηρίζονται έτσι ώστε να αναπτυχθούν σωστά ανεξαρτήτως των εξωτερικών συνθήκων και θα πρέπει ε, να διασφαλιστεί μια συνέχεια στην εκπαίδευση των παιδιών ακόμα και στις πιο δύσκολες των κρίσεων. Ευχαριστώ που αναφερθήκατε στους νέους, στη νεότητα, στη νεολαία όπως θέλετε. Όταν πήγαμε στην Τουρκία, στους καταβλισμούς, ε, αυτή η ηλικιακή κατηγορία είναι το πρόβλημα. Είναι αυτοί που απελπίζονται, είναι αυτοί που θέλουν να φύγουν βλέποντας ότι δεν έχουν μέλλον εκεί και όταν ρωτήσαμε τι διέξοδος υπάρχει για αυτά τα παιδιά, δυστυχώς δεν μας προσφέρθηκαν πολλές απαντήσεις. Δεν μιλάμε για την εκπαίδευση μόνο των παιδιών, αλλά το πώς θα μπορέσουμε. Ε, και κάποιες χώρες έχουν ανοίξει θέσεις σε σχολεία, σε λύκεια, σε γυμνάσια κτλ. Ε, και στη δική μου χώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε νέες προοπτικές. Σας ευχαριστώ όλες σας. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις σας. Ακούσαμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εργαζομένων επιτόπου, Είναι ομαδική η προσπάθεια αυτή την οποία κάνετε και έχει μείνει και λίγος χρόνος για συζήτηση. Θα ξεκινήσω με τον Γκουερέρο, ο οποίος είναι υπεύθυνο και για την διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη και τις ανάγκες οι οποίες αλλάζουν για την ανθρωπιστική βοήθεια στο μέλλον. Καταρχήν, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί με αυτό το σχέδιο ψηφίσματος μπορούμε να μιλήσουμε για την εκπαίδευση Τις ανθρωπιστικές κρίσεις, ε, είτε προκαλούνται από σειράξεις είτε από φυσικές καταστροφές. Γιατί θα πρέπει να ανταποκριθούμε έγκαιρα, γιατί μπορεί να είναι μακροχρόνιες αυτές οι κρίσεις και να διαρκέσουν όσο και η εκπαίδευση μιας γενιάς. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για αριθμητικά στοιχεία, γιατί τα στοιχεία που μας δώσατε ε, είναι χαρακτηριστικά. Αλλά η τελευταία παρέμβασή σας αναφέρθηκε σε επένδυση και όχι δαπάνη. Το αυτό μας είχε και, το, και ο κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στη δεκαετία του 80, δηλαδή ε, ότι μας ενδιαφέρει η ευημερία των ανθρώπων, άρα πρόκειται για επένδυση και όχι για δαπάνη. Στις ανεπτυγμένες χώρες μία κρίση δεν έχει τις ίδιες ε, επιπτώσεις Έχω ασχοληθεί με το τομέα της εκπαίδευσης και είχαμε πει ότι η εκπαίδευση δίνει ζωτική σημασία εχέγγυα στους νέους και καθορίζει το μέλλον τους και επιτρέπει τη συλλογική ανάπτυξη καθώς και κοινωνική και επίσης μειώνονται οι ανισότητες στην κοινωνία. Όταν πρόκειται για καταστάσεις κρίσης, η εκπαίδευση έχει πολλαπλούς στόχους. Καταρχήν προβάλλει την ειρήνη, προαγάει την ειρήνη. Ένα παιδί το οποίο εκπαιδεύεται σε έναν καταβλισμό μέσα στα πλαίσια της ανθρωπιστικής κρίσης στην ουσία είναι ένα στοιχείο υπέρ της ειρήνης και κατά των σειράξεων και επίσης αποσοβεί ορισμένες κρίσεις. Έχουμε την πείρα στο, με το έμπολα και το γεγονός ότι μέσω των παιδιών αντέδρασαν και οι οικογένειες ανταποκρινόμενες στην κρίση αυτή και όσον αφορά την πρόληψη και την μείωση των κινδύνων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, η εκπαίδευση των παιδιών είναι ένα απαράβατο στοιχείο. Η Λίντα αναφέρθηκε στην κατάσταση στους καταβλισμούς στην Τουρκία. Εγώ δύο εβδομάδες πριν στη Συρία και το Λίβανο επισκέφτηκα καταβλισμούς προσφύγων και έχω την ίδια εμπειρία με σας. Δηλαδή οι γονείς των παιδιών είναι διατεθειμένοι να μην τρέφονται καλά προκειμένου να εκπαιδευτούν τα παιδιά τους. Και επίσης το βασικό στοιχείο για να παραμείνουν εκεί ή να μεταφερθούν ε, αλλού με κίνδυνο της ζωής τους. Το στοιχείο, το καταλητικό, είναι το μέλλον των παιδιών τους. Αν θεωρήσουν οι γονείς ότι εκεί όπου βρίσκονται τα παιδιά τους δεν θα έχουν εκπαίδευση για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, τότε θέλουν να διαφύγουν προς άλλες κατευθύνσεις. Δηλαδή είναι διατεθειμένοι να διαπλέψουν τη Μεσόγειο, να την διασχίσουν έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών τους. Η πολιτική μου ομάδα ζήτησε, υπέρ, και τάχθηκε υπέρ της αύξησης των πόρων. Μιλάμε για ένα 26% για την ανθρωπιστική βοήθεια. Θα θέλαμε και το είπαμε στην Επιτροπή αυτή να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό σε αυτό το 4% για την βοήθεια προς την εκπαίδευση και το World Vision θα πρέπει να προωθήσει μια πολυετή, έναν πολυετή προγραμματισμό. Οι επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης δεν μπορούν να είναι βραχυπρόθεσμες. Δεν μπορούν να τεθούν σε ετήσια βάση, διότι ο εκπαιδευτικός κύκλος διαρκεί κανονικά 5 με 10 χρόνια. Αυτό είναι το ελάχιστο. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει πολυετής ε, προγραμματισμός. Αύριο θα μιλήσουμε και για την ε, δική μου έκθεση μέσα στα πλαίσια της ε, παγκόσμιας διάσκεψης έτσι ώστε να υπάρξει ένα παγκόσμιο ταμείο για την ανθρωπιστική βοήθεια για να, προωθηθεί να προωθούν οι χορηγίες για την εκπαίδευση και η χρηματοδότησή της. Όσοι φεύγουν από έναν πόλεμο γνωρίζουν ότι με την εκπαίδευση οι ίδιοι δεν θα συμμετέχουν στο επόμενο στάδιο του ιδίου πολέμου. Αν λοιπόν έχουν μία ποιοτική εκπαίδευση με βάση τις αξίες της συνεργασίας, ίσως να μην παρατωθούν και οι πόλεμοι. Ευχαριστούμε Ρίκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω για την Ρή και να ευχαριστήσω και τι άλλε ομάδες που υποστήριξαν τη συμπερίληψη του θέματο αυτό στην ημερήσια διάταξη και όχι μόνο για την Επιτροπή μα, αλλά και για την Ολομέλεια μάλιστα. Με την ερώτησή σα νομίζω ότι τίθεται το θέμα τη ευαισθητοποίηση για την ανάγκη για εκπαίδευση σε περιστάσει και περιπτώσει κρίσεων αλλά και σε το θέμα του ποσοστού που διαθέτουμε για την εκπαίδευση και υπό την έννοια αυτή καλωσορίζω ασφόλως την ανακοίνωση του και την δήλωση του Επιτρόπου Στυλιανίδη. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να συζητήσουμε τα όσα συμβαίνουν ήδη και να θέσουμε το θέμα μεταξύ της εκπαίδευσης ε, σε περιπτώσεις κατεπίγουσης ανάγκης και της εκπαίδευσης σε καταστάσεις μετανάστασης. Αυτό θα το μετωπίσουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέσσερις ερωτήσεις έχω να θέσω. Σύντομα. Προκειμένου να μπορέσουμε να ακούσουμε και απαρκώς τις απαντήσεις τεκμηριωμένες. Καταρχάς, αυτή η αύξηση 2-4% τι αντίκτυπο θα έχει. Πόσα παιδιά προσπαθούμε να αγγίξουμε εδώ πέρα. Έχουμε τα αριθμητικά στοιχεία των παιδιών που δεν πηγαίνουν σχολείο. Υπάρχει οποιαδήποτε εκτίμηση για το πόσα παιδιά θα μπορέσουμε να... σε πόσα παιδιά παραπάνω θα μπορέσουμε να δώσουμε εκπαίδευση. Δεύτερο θέμα, το θέμα συντονισμού. Το είπε η πρόεδρος αυτό και κατά πάσα πιθανότητα η επικεφαλής της UNICEF θα μπορέσει να μας απαντήσει. Γιατί υπάρχουν τόσες ε, πολλές πρωτοβουλίες. Global Business Initiative για την εκπαίδευση κτλ. Και φυσικά πάντα ανακύπτει το προφανές ερώτημα. Τα χρήματα αυτά τελικά καταλήγουν σε όσους τα χρειάζονται ή μήπως τελικά έχουμε τόσους ενδιάμεσους που δεν φτάνουν στον τελικό προορισμό τους τα χρήματα αυτά. Πείτε μας και λόγια λοιπόν και γι' αυτό και για το συντονισμό των δράσεων στην διεθνή κοινότητα. Τρίτο σημείο. Συμπεριλαμβάνουμε αρκετά πράγματα σε διαφορά αφορά το έργο μας τόπου. Η εμπειρία της ε, διευθύντριας της UNICEF από το Κωσυφοπέδιο θα χρησιμεύσει σίγουρα για να απαντήσουμε την ερώτηση αυτή. Θυμάμαι ότι υπήρχε ένα ανεπίσημο άτυπο σύστημα υπό, τον, υπό τους Σέρβους. Υπήρχε αυτό το σύστημα. Και πρόσφατα μίλησα με εκπρόσωπο από τη Συρία και νημαυρίστηκε. Είπε ότι δεν ήρθαν καν σε επαφή μαζί του και ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να πληρωθούν όλα τα διεθνή κριτηρία για τη βοήθεια τα οποία ήθελε. Επιτόπου λοιπόν κάνουν καλή δουλειά σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση σε περιοχές κρίσης. Έχουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα επαρκούς συμπερίληψης όλων των παραγόντων. Μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Τέλος. Ε, τελευταία ερώτηση. Η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και θέσεων εργασίας. Ε, ιδιαίτερα για τους εφήβους. πώς μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα, αυτές τις ικανότητες αν δεν έχουν δουλειά. Ε, η εκπαίδευση αποτελεί κίνητρο μετανάστευση τελική ανάλυση. Υπάρχει κάποια μακροπρόθεσμη στρατηγική για αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ελίντα, muchísimas gracias a, a todas las ponentes de hoy por Ευχαριστώ πολύ όλες ε, τις ε, εκπροσώπους για τα πολύ ενδιαφέροντα μηνύματά τους και νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι ύψης της ε, σημασίας όχι μόνο για την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα και για τα παιδιά, τα εκτοπισμένα παιδιά τα οποία βρίσκονται τώρα σε προσφυγικούς καταβλισμούς αλλά γιατί επί της ουσίας θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά ε, είναι ότι θα πρέπει να άρουμε τα προσκόμματα μεταξύ αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Στην ουσία αυτό το πρόσκομα δεν υπάρχει και το βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτό το, ε, αυτή η ερώτηση έχει και ένα επιπρόσθετο στοιχείο θα θέλαμε να φτάσουμε στο στόχο της Ατζέντα 2030 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και γνωρίζουμε τη διάδραση που, υπάρχουν, που υπάρχει μεταξύ αυτών των στόχων. Δηλαδή μιλάμε για ποιοτική εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και ισότητα των δύο φύλων. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση και να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση για την εκπαίδευση πέρα από τις ε, κρίσεις ε, και ε, την επίγουσα ανάγκη. Διότι μιλάμε για ε, διεύρυνση του, του ποσοστού αυτού και μιλάμε και για διπλασιασμό από 2 σε 4% του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτές οι πρωτοβουλίες θίγουν πραγματικά το θέμα της χρηματοδότησης. Δεν θα ήταν καλύτερα να υπάρχει ένα παγκόσμιο ταμείο για την εκπαίδευση. Αυτό λέχθη στη διάσκεψη κορυφής της ε, Νέας Υόρκης. Δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα παγκόσμιο ταμείο για να αντιμετωπίσουμε τη φυματίωση, την ελονοσία και ούτω καθεξής. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει σωστή διαχείριση με εμπειρογνώμονες σε επίπεδο κυβερνήσεων και θεσμικών οργάνων. Όπως είπαν και οι εκπρόσωποι, αυτό που έχει σημασία είναι η φυσική και ψυχολογική προστασία του παιδιού. Γι' αυτό χρειάζονται ασφαλή σημεία διδασκαλίας και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέσουμε τους κατάλληλους πόρους για να μπορούμε να προστατεύσουμε τα σχολεία και τα πανεπιστήμια σε περίπτωση σύρξης. Επειδή έχει σημασία να ακούσουμε εσάς περισσότερο και όχι εμάς, θα ήθελα να μου πείτε πώς μπορεί να οριστεί αυτό το Παγκόσμιο Ταμείο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι τις επίγουσες ε, ανάγκες και τι σκέφτεστε μέχρι το 2030 για αυτή την πρόταση. Εκτός Τώρα ναι, τώρα σας ακούμε πάρα πολύ μια τέλουσα συζήτηση αυτή που κάνουμε. Θα ήθελα να πω μόνο στους προσκεκλημένους μου ότι καταρτίζω μια έκθεση που περνάει ε, από τα κοινοβούλια για τον ιδιωτικό κλάδο και την ανάπτυξη. Αν πάει λοιπόν στην... Ε, θα πάει στην Ολομέλεια στην τέλη του έτους. Το όλο θέμα της εκπαίδευση, αν το δούμε από ολιστικής ε, άποψης, θα πρέπει να δούμε ποιος απασχολεί τελικά την πλειοψηφία του κόσμου που εκπαιδεύεται. Δεν είναι κρατική φορή, είναι ο δυτικό κλάδο. Οι δουλειέ στον δυτικό κλάδο γεννιούνται. Η εκπαίδευση λοιπόν καθίσταται η υπηρεσία. Η υπηρεσία προ τον δυτικό κλάδο. Στη δική μα νοοτροπία ωστόσο. Ε, εμπλέκουμε τον δυτικό κλάδο, ιδιαίτερα στι αναπτυξιόμενε χώρε σε ό,τι αφορά την παροχή εκπαίδευση, βλέπουμε τον ε, δυτικό κλάδο ω κάτι ξεχωριστό, αντιλώ από την πραγματική οικονομία των χωρών. Αλλά αν κάνουμε μια ανάλυση σε κάθε, σε κάθε αναπτυσσόμενη χώρα, πού είναι οι δουλειές, και όλα τα μάντρα του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, τη παγκοσμία, τράπεζα, τι λένε, να μειώσουμε την απασχόληση στο δημόσιο τομέα και να αυξηθούν οι δουλειέ στον ειδικό κλάδο. Είτε μιλάμε για ορυχεία, είτε μιλάμε παροχή υπηρεσιών, για παροχή υπηρεσιών, είτε μιλάμε για την Αφρική, είτε μιλάμε για το Βιετνάμ. Ο ιδιωτικό κλάδο είναι αυτό που τελικά χρησιμοποιεί τα άτομα αυτά τα οποία έχουν εκπαίδευση και όπως στη Σιλάνκα θα δείτε ότι ο δημόσιος τομέας τελικά καταλήγει με τους λιγότερο εκπαιδευμένους. Τι ήθελα να πω στην τελική ανάλυση. Γιατί δεν απαιτούμε πιο πολύ συμμετοχή και πιο πολλά από τον ιδιωτικό κλάδο, γιατί όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται για να εξυπηρετήσει τελικά τον ιδιωτικό κλάδο. Αλλά δεν του ζητάμε τίποτα να συνδράμει στην εκπαίδευση. Ο φορολογούμενο τελικά πρέπει να τα πληρώνει όλα. Και ο ιδιωτικό κλάδο τίποτα. Ε, ιδιαίτερα οι διεθνεί ε, όμιλοι που δεν πληρώνουν και φόρους πουθενά και σήμερα ακούσαμε ότι το Facebook η πιο υψηλή αξία στην εταιρεία του κόσμου πληρώνει λιγότερου φόρου από ότι... Τι να σας πω ένα κανονικό φορολογούμενο στη Βρετανία. Και τι ζητάμε από τη Facebook να κάνει όμω για την εκπαίδευση. Βοηθάει καθόλου τι αναπτυσσόμενε χώρε στην εκπαίδευση. Από την GK, η Tengelog και από άλλε εταιρείε. Έχει συμμετάσχει κανεί πουθενά. Όχι. Πουθενά. Και γιατί. Σας ευχαριστώ. Ε, ας ξεκινήσουμε να πληρώνουν τους φόρους τους τουλάχιστον, λέει η Πρόεδρος. Θα βοηθούσε και αυτό. Μαρία Χόιμπροκ και η κυρία Χάουταλα μετά. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι δύο πράγματα μας κάνουν εντύπωση και στις παρουσιάσεις και στη συζήτηση και θα πρέπει να τα αντιληφθούμε. Είναι η παρατεταμένη διάρκεια των συγκρούσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι καταβλισμοί μεταναστών ε, τελικά καταλήγουν να φιλοξενούν άτομα ε, για 20 χρόνια και παραπάνω, όπως γίνεται με του Ομαλούς στην Κένια. Και αν θέλουμε να υπάρχει μια οποιοδήποτε ελπίδα ζωής μετά τον καταβλισμό, θα πρέπει να υπάρχει και μια γέφυρα επιστροφής θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν εκπαίδευση και να υπάρχει σε διάφορα επίπεδα του πληθυσμού για όλες τις γενιές. Θα ήθελα λίγο παραπάνω έμφαση ενδεχομένω στην κατάσταση των καταβλισμών των μεταναστών. Γι' αυτό λοιπόν θα καταρτήσουμε και κάποιες τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Και αυτό γιατί ε, δεν βλέπω πουθενά να αναφέρεται ρητά το θέμα αυτό. Το δεύτερο θέμα που έχω αναφέρω κατανοούμε και αυτό περιλαμβάνεται πολύ καλά στο σχέδιο ψηφίσματος ότι τα ευάλωτα κράτη πραγματικά πλήττονται σε ό,τι αφορά την έλλειψη χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, και για όσο διαφορά τις γενιές ολόκληρες που χάνονται από τον κύκλο εκπαίδευσης. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τη Διεθνή Εταιρική Σχέση για την Εκπαίδευση. Πρόκειται για μια οργάνωση που πραγματικά υποστηρίζει την ε, δημιουργία σωστών εκπαιδευτικών συστημάτων στη χώρα. Και πραγματικά αξίζει να επενδύσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Και είδα και σε μία από τις παρουσιάσεις ότι αυτό το Global Partnership for Education μπορεί να κινητοποιήσει και πάρα πολύ γρήγορες δράσεις σε περιπτώσεις κατεπίγουσες ανάγκης. Αν ρωτιέμαι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συνεργαστεί λίγο παραπάνω για να δώσει όθηση στο διεθνή διάλογο σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση ειρήνης και κρατών, το G7+, για τα ευάλωτα κράτη, όπως ονομάζεται. Γιατί τι βλέπουμε, ότι ακόμα και οι στόχοι της χιλιετίας ότι βάζει την ανάπτυξη δεν έχουν επιτευχθεί στα ευάλωτα κράτη λόγω κατάρρευσης και του κράτους και των δομών και ίσως λοιπόν ο κλάδος της εκπαίδευσης θα μπορούσε να τονιστεί λίγο γιατί βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε εταιρική σχέση για παράδειγμα με τον Νότιο Σουδάν. Το Νότιο Σουδάν αναφέρθηκε από τους ομιλητές. Γιατί να μην προσπαθήσουμε λοιπόν να αφιερώσουμε πιο πολλούς πόρους για πιο πολλά αποτελέσματα για τέτοιες καταστάσεις. Συμφωνώ απόλυτα με τον ομιλητή που είπε ότι ο τίτλος ε, θα έπρεπε να είναι η εκπαίδευση των παιδιών σε κατατήρους ανάγκες και σε παρτιναμένες περιπτώσεις κρίσεων, γιατί αυτό ισχύει σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς. Αναφέρθηκε επίσης ότι η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση στην κοινωνία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες και τα κορίτσια. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα κατανοήσουμε καλύτερα. Μεταξύ άλλων το γεγονός ότι η εκπαίδευση υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών. Η Αντζελίνα Τζολί είδα ότι χρηματοδοτεί ένα ε, σχολείο κοντά στην Μακάνη στην Κένια ε, ένα σχολείο εσωτερικό, στο για κορίτσια. Είναι έξυπνη ιδέα αυτή, γιατί τα κορίτσια έτσι δεν είναι στα χέρια των γονιών τους, που ενδεχομένω ε, δεν θα εξαναγκάσουν να παντρευτούν και έτσι έχουν την εκπαίδευση που χρειάζονται. Νομίζω ότι χρειάζονται λοιπόν πιο πολλές ε, πρωτοβουλίε τέτοιων ειδών. Μαρία Χόιμπρουκ και ο, ε, μετά ο Χουάκιμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την επισκόπηση που μας δώσατε για την κατάσταση στην εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και φυσικά καλωσορίζουμε το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός αυξάνεται σε 4% αλλά παρόλα αυτά διαπιστώνουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο κενό χάσμα στη χρηματοδότηση αυτών των στοιχείων. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν επιπρόσθετοι πόροι, γιατί οι κρίσει πολλαπλασιάζονται, δεν μειώνονται. Και τα άτομα που ζουν σε τέτοιους καταβλισμού αυξάνονται. Αυτό λοιπόν επιτάσσει την κινητοποίηση μεγαλύτερων πόρων. Και αν δεν φτάνει ο τομέα ε, της ε, υγείας ε, και της, της, του επιστησμού θα πρέπει να κοιτάξουμε για την κλάδα αυτό. Ανησυχώ λοιπόν ιδιαίτερα για το θέμα της χρηματοδότησης Και η κυρία Λορέντσο ανέφερε τα αριθμητικά στοιχεία. Είπατε ότι αυξήθηκε η χρηματοδότηση. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, είναι ασφαλής αυτή η χρηματοδότηση, έχει περιληφθεί στον προπολογισμό, μπορούν να δαπανηθούν αυτά τα κονδύλια, ή μήπω υπάρχουν τέτοιε επικεφαλίδε χωρί να υπάρχει η μήπως υπαρχουν τετοιε επικεφαλίτε χωρι Πιστεύω ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Από τις παρουσιάσεις ε, των εμπειρογνωμόνων προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα χρηματοδότησης αμυγός. Φυσικά υπάρχει και, υπάρχουν και κονδύλια, αλλά δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η χρήση των πόλων δεν γίνεται με στοχευμένο τρόπο και έτσι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές αρμοδιότητες, υπάρχουν θέματα συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, η αναπτυξιακή πολιτική βασίζεται στις ε, Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα τα κράτη-μέλη ακολουθούν δική τους πολιτική σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Υπάρχουν ειδικά ταμεία όπως το Ταμείο για την Ανάπτυξη, τα οποία δεν αποτελούν καν τμήμα του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού αλλά απλά ένα από ένα διοικητικό όργανο να καθορίζεται. Ε, στο σημείο αυτό θεωρώ ότι και θα πρέπει να κάτσουμε να κοιτάξουμε και να δούμε, όπως είπε και η Πρόεδρος. Και όπως προεκύψε σε επίσκεψη στην Τουρκία για τους πρόσφυγες από τη Συρία, δεν φτάνει μόνο ο άρτος ε, για να ζήσει ο άνθρωπος, ε, όπως λέει και η βίβλος. Το θέμα είναι και πώς θα προετοιμαστεί η νέα γενιά για το μέλλον, πώς θα την προετοιμάσουμε εμείς. Αυτό είναι το επόμενο σημείο και νομίζω ότι η εκπαίδευση αποτελεί κατεξοχήν αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε κράτους. Είναι κρατική ευθύνη η προετοιμασία της κάθε γενιάς για το μέλλον. Τι γίνεται λοιπόν σε κράτη που δεν αντιλαμβάνονται αυτή την ευθύνη όπου οι γονεί ε, δεν στέλνουν καν τα παιδιά του στο σχολείο ή ενδεχομένω τα βγάζουν από το σχολείο γιατί χρειάζονται τα εργατικά χέρια του. Και πρέπει να συνδράμουν στην οικογένεια. Εδώ νομίζω ότι τίθεται και ένα πολιτικό ζήτημα. Το όνομα του Σουδάν ήδη αναφέρθηκε ως παράδειγμα. Εγώ παρευρέθηκα εκεί και μίλησα με αναπτυξιακούς ε, ε, βοηθούς και είχαν χρήματα να χτίσουν σχολεία. Αυτό που δεν είχαν όμως ήταν χρήματα να προσλάβουν δασκάλους. Και όταν ε, ρώτησαν τους τοπικούς άρχοντες κατά πόσον ε, μπορούσαν να διαθέσουν χρήματα για να προσλάβουν ένα δάσκαλο, η απάντηση ήταν «Μα εμείς χτίσαμε τα σχολεία». Και πάνω από το 90% του προϋπολογισμού του Νοτίου Σοδάν δαπανάται σε στρατιωτικές δαπάνες. Θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε την πολιτική πίεση επί που πιστεύω αν εμείς συνεργαζόμαστε και αυτοί να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Ναι, με, λοιπόν να υπάρχει υποστήριξη, αλλά να χρησιμοποιείται στοχευμένα. Για τα άτομα τα οποία διώκονται στα, στους καταβλισμούς υπάρχει μια κάποια δομή την οποία μπορούμε να επηρεάσουμε, αλλά λίγοι είναι σε καταβλισμούς. Στην Νότια Τουρκία για παράδειγμα, οι Σύριοι πρόσφυγες μόνο κατά 12-13% ζουν σε τέτοια καταλήμματα, σε καταβλισμού. Οι πιο πολλοί βρίσκονται σε χωριά, έξω τα χωριά και εδώ παρουσιάζεται το μεγάλο πρόβλημα γιατί μιλάμε για χρόνια πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη γενιά η οποία δεν εκπαιδεύεται όχι μόνο παιδιά αλλά και οι νέοι όπως είπε και η Πρόεδρος. Ως εκ τούτου πιστεύω. Και έτσι ερμηνεύω και το ψήφισμα βάσει της προφορικής ερώτησης. Αυτά τα θέματα θα πρέπει να επισημάνουμε. Καταρχάς, ε, ότι στην αναπτυξική βοήθεια το σκέλος της εκπαίδευσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με προτεραιότητα και να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των μεμονωμένων φορέων και να κοιτάξουμε και τις, ε, την πολιτική πίεση στις χώρες εκείνες που χρειάζονται υποστήριξη προκειμένου πραγματικά να αποτελέσει σημείο προτεραιότητας διεκπαίδευσης και στις χώρες αυτές. Um, Ευχαριστώ σε όσους πήραν το λόγο. Έλαβα κάποιες πληροφορίες ε, <clears throat> για την παρουσία και άλλων οργανώσεων που είναι δραστήριες για τα παιδιά σε κατεπίγουσες καταστάσεις. Η Ούρα, σαν παράδειγμα, που ασχολείται με την Συρία, έκαναν μια παρουσίαση ε, στο Κοινοβούλιο για τις απαράδεκτες συνθήκες με τις οποίες δραστηριοποιούνται η οργάνωση Save the Children, η οργάνωση Children in Crisis. Κάποιοι από εσά είστε εδώ και προσπαθείτε να φέρετε θετικές αλλαγές έχουν τεθεί πολλές ερωτήσεις. Να θέσω και εγώ κάποιες προς την Επιτροπή. Χρήματα και για τους νέους, όχι μόνο για τα παιδιά. 20-23 23 ετών. Τι δυνατότητες υπάρχουν. Και πώς στηρίζουμε τις χώρες αυτές. Βοηθάμε τις κυβερνήσεις που υποδέχονται ε, στα δικά του συστήματα. Στην Τουρκία είδαμε ας πούμε ότι υπήρχαν διπλές βάρδιες στα τουρκικά σχολεία για να βολέψουν τα παιδιά των προσφύγων. Τι κάνουμε για να βοηθήσουμε τις χώρες που υποδέχονται τους πρόσφυγες και τι γίνεται ε, για την εργασία των καθηγητών και των δασκάλων από τις χώρες διαφυγής. Η UNICEF ε, ε, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τους ανθρώπους αυτούς αλλά θα ήθελα να πληρώνονται καλύτερα και με πιο τακτικό τρόπο. Είναι περίπλοκα θέματα αυτά βέβαια. Δεν ξέρω ποια από όλες θα ήθελα. Ίσως ο, η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα. Κυρία Λορέντσο πρώτα μάλλον. Να ξεκινήσω με τα υπόλοιπα θέματα τρία σημεία. Το πρώτο αφορά τη χρηματοδότηση σε σχέση με τις πιστώσεις ελεγχόμενη από τον συνάδελφο της ΕΚΟ να πω ότι αν αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια από 2 σε 4% δεν λύνει στο πρόβλημα των πολιετών προγραμμάτων ποιος είναι αυτός ο οποίος χρηματοδοτεί ε, και σε ποιο βαθμό τα χρήματα αυτά προέρχονται από, τα αναπτυξιακά, από τις αναπτυξιακές πιστώσεις. Η αριθμή που σας παρουσίασα δείχνει ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα πράγματα για κάθε μία από τις κατηγορίες τις οποίες δραστηριοποιούμε. Από το 2014 μέχρι το 2020 θα δαπανίσουμε 1,7 δις σε εύθραυστες χώρες. Τα ποσά αυτά είναι διαθέσιμα, είναι ασφαλισμένα. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν στην ενδιάμεση αναθεώρηση βέβαια. Για λόγους κυρίως μη απορρόφησης. Το πρόβλημα είναι ότι σε πολλές από τις χώρες αυτές αυτό είναι το πρόβλημα. Οι εύθραυστες χώρες έχουν χαμηλά επίπεδα θεσμικής λειτουργίας και αν τους δίνουμε περισσότερα χρήματα δεν πετυχαίνουμε περισσότερα αποτελέσματα Πρέπει να ενισχύουμε την δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων ε, και έχουμε τεράστια προβλήματα απορροφητικότητας. Και εδώ βρισκόμαστε στη φάση της απορρόφησης και εδώ ε, έχουμε προβλήματα. Η εφαρμογή είναι κάτι που δεν ε, ενδιαφέρει φαίνεται κανέναν. Όλοι μιλάνε για τη χρηματοδότηση αλλά δεν μιλάνε για τη διαχειριστική ικανότητα, την, την ελεγκτική ικανότητα. Όσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση, τόσο περισσότερη οργάνωση χρειάζεται. Και όσο πιο εύθραυστη είναι η κατάσταση, τόσο λιγότερος ανθρώπους έχει στη διάθεσή σου. Το θέμα των εύθραστων χωρών είναι πρόβλημα στην εκπαίδευση. Έχουμε ε, τη UNICEF, τη UNICEF και κανέναν άλλο που να ασχολείται με τα θέματα οργάνωσης της εκπαίδευσης. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω, ίσως το αντιμετωπίζουν και οι αντίστοιχε υπηρεσίε των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε τεράστια προβλήματα για προσλήψεις καθηγητών, στελεχών, η κατάσταση είναι περίπλοκη. Και έρχομαι στο τρίτο θέμα που αφορά το Παγκόσμιο Ταμείο. Προσωπικά και προσωπώντας την οργάνωση το ταμείο δεν είναι η λύση. Ένα τέτοιο ταμείο θα οδηγήσει στην πολυδιάσπαση του τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει έτσι και αλλιώς το Global Partnership για την εκπαίδευση. Ας προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε αυτό το καταπίστευμα απαιτείται περισσότερη δυνατότητα και εκτελεστική δράση από μέρους του, αλλά δυστυχώς υποχρηματοδοτείται ιδιαιτέρως. Πήρε τα μισά από αυτά τα οποία είχε ζητήσει, πήρε 3,5 δις. Οπότε γιατί να δημιουργήσουμε ένα νέο διεθνές ταμείο. Η διαχείριση για να μπορέσει να είναι αποτελεσματική απαιτεί 10 χρόνια, ας που να καταστεί κάτι τέτοιο λειτουργικό. Έχουμε ένα τέτοιο ταμείο το οποίο υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια, μπορούμε να το ενισχύσουμε για να λειτουργήσει σωστά. Ήδη δουλεύει κατά το ίμιση σε εύθραυστες χώρες, ευαίσθητες χώρες. Για τις δύο τελευταίες σας ερωτήσεις, για τα καταπιστεύματα, για, τα ταμεία μάλλον, για την νεότητα. Ε, υπάρχουν πολλές χώρες τις οποίες εργαζόμαστε, οι μισές από αυτές γύρω στις 22-23 έχουν συστατικά της επαγγελματικής κατάρτισης. Δυστυχώς όμως η επαγγελματική κατάρτιση συνδέεται με το επίπεδο αν θέλετε των κυβερνητικών διοικητικών ικανοτήτων και το επίπεδο της ανάπτυξης του δημόσιου τομέα και της σχέσεις με την εκπαίδευση και την ανεργία. Όσο πιο έθραστη είναι μια χώρα τόσο πιο δύσκολο είναι να υπάρξει παρέμβαση στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Και τέλος, είπα αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να προγραμματίζει κανείς σε επίπεδο χώρας. Σε ορισμένες χώρες μπορέσαμε να στηρίξουμε τα κυβερνητικά συστήματα και να στηρίξουμε ακριβώς τις διοικητικές δομές να εντάξουν τους πρόσφυγες. Σε άλλες χώρες δεν γίνεται κάτι τέτοιο, η πολιτική της χώρας δεν μας το επιτρέπει, οπότε δημιουργούμε εμείς παράλληλα αυτόνομα συστήματα τα οποία γίνονται αντικείμενο διαχείρισης από τις ΜΚΟ. Τέλος. Έχουμε μία συγκεκριμένη πίστοση 60 εκατομμυρίων για τα επόμενα 6 χρόνια για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της έφτραστης χώρες και το πρώτο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτών, δηλαδή των δασκάλων, που είναι ακατάλληλοι μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις η κυρία Λένσου που έθεσε ο κύριος Στήρ. Κατά πόσο θα αυξηθεί ε, ο αριθμός των ανθρώπων που βοηθούμε με, με την αύξηση αυτή 4%. Έχουμε 23 δις που θα έχουμε δαπανίσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Συνολικά θα έχουμε φτάσει σε 1,5 εκατομμύριο παιδιά σε 26 χώρες. Αυτό εξαρτάται βέβαια πλήρως από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι προτάσεις για τα διάφορα προγράμματα. Η συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και με την Ερυθρά Ημισέλινο και τον Ερυθρό Σταυρό. Έχουμε λοιπόν διάφορα προγράμματα τα οποία ε, καλύπτουν ε, ε, μικρούς αριθμούς ανθρώπων σε βάθος και ευρύτερα προγράμματα τα οποία με πιο αν θέλετε επιδερμικό τρόπο καλύπτουν όμως ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Λοιπόν, ε, υπάρχουν πολλές προκλήσεις τις οποίες πρέπει να καλύψουμε και εξαρτάται με ποιο τρόπο θα ε, στοχεύσουμε. Για τη δεύτερη ερώτηση, ότι υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες και ο συντονισμός όπως είπε και η συνάδελφος είναι ένα ξεκάθαρο θέμα. Θεωρούμε ότι είναι βασικό αυτό και θα πρέπει εμείς να ελαχιστοποιήσουμε ε, το κόστος των συναλλάκων τότε μόνο θα έχει νόημα αυτό το οποίο κάνουμε. Το θέμα είναι πώς το κάνεις αυτό, πώς σταματάς τους ανθρώπους να ξεκινήσουν νέες πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω αν έχουμε εκπροσώπους από τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά πράγματι σε ποιο βαθμό μπορεί ε, ο οργανισμός αυτός να λειτουργήσει συντονιστικά και πώς μπορούμε να προσελκύσουμε και τον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να το αντικείμενο ε, συντονισμού. Εφόσον έχουμε ένα διεθνές ταμείο το οποίο είναι υποχρηματοδοτούμενο, γιατί να δημιουργηθεί κι άλλο ένα. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ε, Έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα για την εκπαίδευση και την επιρροή τους στην οικογενειακή ζωή. Όλα αυτά εξελίσσονται συνεχώς. Όλες οι ικανότητες που μπορεί να βοηθήσουν τους νέους να αποδώσουν περισσότερο πρέπει να στηριχθούν. Πρέπει να κατανοήσουμε τι ζήτηση υπάρχει εγώ έχω εργαστεί σε θέματα επαγγελματικής κατάρτασης, έχουμε προχωρήσει στην παραγωγή ραπτών, φουρνάριδων κτλ. Πρέπει να ξέρουμε τις ανάγκες λοιπόν, γιατί αλλιώς θα αποτύχουμε και ε, στην ουσία τους προετοιμάζουμε και αυτούς να αποφύγουν και πραγματικά είναι τρομερό το πόσο επικίνδυνο μάλιστα τρομακτικό είναι μια ομάδα νέων απογοητευμένων χωρίς την αίσθηση του μέλλοντος. Υπήρξαν επίσης ε, ε, και κάποια προγράμματα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες χωρών πριν την ανεξαρτησία και αμέσως μετά. Νομίζω ότι ό,τι κέρδη είχαμε στον τομέα της εκπαίδευσης, τα παραδείγματα που έχουμε μας δείχνουν ότι απέτυχαν δυστυχώς. Στην ουσία ο κουβάς είχε μία τρύπα, το βαρέλι είχε μία τρύπα, δίναμε εμείς αλλά χανόντουσαν τα χρήματα. Η εκπαίδευση είναι ένα κομμάτι μιας ευρύτερης δομής και αυτό καθιστά το σύστημα περίπλοκο. Και αυτό είδαμε στο Νότιο Σουδάν. Είδαμε πόσο γρήγορα εξελίχθηκαν τα πράγματα και σε ποιο βαθμό και με πόσο τρομερή ταχύτητα το Υπουργείο Παιδείας στην περιοχή του Άνω Νείλου στην ουσία διαλύθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Από τις μεγαλύτερες ε, επιτυχίες είναι ας πούμε να συμπεριλάβουμε και τις απόψεις ε, των γονέων που κατανοούν τι σημασία έχει η εκπαίδευση. Τα οικοτροφία είναι πολύ ακριβά, ε, δουλεύουν καλά αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να πείσουμε τους γονείς εδώ ότι πρέπει να στέλνουν τα παιδιά τους. Εκπαιδεύουμε και τους γονείς. Είχαμε επίσης Επιτυχίες σημαντικές στο Βόρειο Ιράκ με τους ενήλικες, με τους υπεύθυνους, τους κηδεμόνες μάλλον των οικογενειών. Λοιπόν, έχουμε προχωρήσει και σε περιοχές όπως ο Λίβανος, η Ιορδανία. Ε, έχουμε μιλήσει για τις αστικές περιοχές, έχουμε εκτοπιστέντες πληθυσμούς, με τα παιδιά στο κέντρο των πόλεμων, έχουμε δάσεις, έχουμε δυνατότητα απορρόφησης ενός εκπαιδευτικού συστήματος που έχει προβλήματα να εκπαιδεύσει τα δικά του παιδιά, πόσο μάλλον τα παιδιά των εκτοπισμένων πληθυσμών. Έχουμε προβλήματα με τριπλές βάρδιες, τετραπλές βάρδιες, απίσχναση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η κατάσταση χειροτερεύει. Εγώ είμαι δασκάλα και στην ουσία ναι μεν βοηθάμε τους δάσκαλους, συνεργαζόμαστε μαζί τους για να ελέγξουν όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά φοβάμαι ότι έχουμε μεγάλες απώλειες, οι ΜΚΟ κατηγορούνται ότι απορροφούν πολλούς εκπαιδευτικούς γιατί δίνουν καλύτερες αμοιβέ και τους χρειάζονται εκεί. Πρέπει λοιπόν εμείς να αξιολογήσουμε σωστά, να εκτιμήσουμε, να βοηθήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους δασκάλους γιατί εξαρτώμεθα από τους δασκάλους για να δώσουμε ποιότητα στα μαθήματα. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δοθούν απαντήσεις. Ε, για να ξεκινήσω από το Λίβανο και την πρόσφατη επίσκεψή σας, μία από τις εταιρικές σχέσεις που προωθήσαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και αυτή. Δηλαδή ε, όταν μετακινούνται άνθρωποι στο Λίβανο πάνε στις πιο φτωχές και ευάλωτες περιοχές. Άρα τα προγράμματα μας δεν υποστηρίζουν μόνο τους πρόσφυγες αλλά σχετίζονται με την ανάπτυξη των πιο φτωχών λιβανέζικων κοινοτήτων μέσα στα πλαίσια της ε, κοινωνικής ε, συνοχής. Και αυτό έπρεπε να γίνει ακόμα και πριν από την ε, κρίση σε αυτές τις ε, αποτρόπες καταστάσεις ε, βλέπουμε ότι ευτυχώς ανοίγει ένας πολιτικός δρόμος για να ε, υπάρχει ένα μέλλον για τα παιδιά. Και στο Κωσυφοπέδιο υπήρχε ένα παράλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης και μόνο με το τέλος του πολέμου έγινε λόγος για ενοποιημένο σύστημα εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια μεγάλη ηρωνία ε, που αφορά αυτούς τους τομείς σε σχέση ιδιαίτερα με την ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτό που έχει σημασία είναι ο συντονισμός αποκλειστικά με την πληθώρα πρωτοβουλειών έχουμε μεγάλα χάσματα στη χρηματοδότηση και την εφαρμογή. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και στους δύο τομείς είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι. Ε, επιτόπια υπάρχει και η προσέγγιση των ε, κοινών σημείων, των σημείων διεπαφής ε, και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς μπορούμε να ε, συντονίσουμε την κατάσταση σε σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη. Θεωρούμε ότι έχει μεγάλη σημασία να λάβουμε υπόψη αυτές τις πρωτοβουλίες, αλλά πρέπει να είναι συνεκτικές και συντονισμένες. Είχαμε ε, εξαιρετική συζήτηση. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει συνοχή και η συνεργασία και να μην προσθέσουμε και άλλες πρωτοβουλίες εμείς. Πρέπει να προσθεθούμε σε αυτές που ήδη υπάρχουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τέσσερις ομιλήτριες και να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι η προθεσμία είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, στις 10 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε. Προθεσμία για μεθαύριο για υποβολή ε, τροπολογιών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay. So, um, in fact that Άρα προχωράμε στο επόμενο θέμα που αφορά την απαστολή πραγματογνωμοσύνης Επιτροπής Ανάπτυξης στη Γκάζιεντεπ, στη νότια Τουρκία. Ήταν πολύ μικρή αντιπροσωπεία. Εγώ, ο Ζωακίμ Ζέλ και ο Νόρπερτ Νόιζερ. Ένα μήνα πριν πήγαμε στη Νότια Τουρκία, ε, οργανώσαμε την αποστολή αρκετούς μήνες πριν, πριν γίνει λόγος για την κρίση στην Τουρκία. Έχετε την έκθεση μπροστά σας, μπορείτε να τη διαβάσετε, αλλά να σας πω ορισμένα στοιχεία μόνο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ζουν σε καταβλισμούς. Μόνο το 15% των προσφύγων ζουν σε καταβλισμούς. Το 1,9% των προσφύγων, το 1,9 εκατομμύρια με συγχωρείτε, ζουν ε, σε, στην κοινότητα, έχουν ενταχθεί στις κοινότητες, στις τοπικές κοινότητες. Η κατάσταση, αν ε, λάβουμε υπόψη, σημαίνει τώρα στην Τουρκία, το σκεφτόμουν το Σαββατοκύριακο, η κατάσταση θα οδηγήσει και άλλους να φύγουν από εκεί. Μιλήσαμε με όλους τους ε, φορείς ε, και θα πρέπει να πούμε ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει δαπανίσει πολλά χρήματα και χρόνο για να υποστηρίξει τους ε, πρόσφυγες και να τους ενσωματώσει αυτούς τους προσφύγους από το Ιράκ, το Αφγανιστάν, αλλά κυρίως από τη Συρία. Οι ίδιοι οι καταβλισμοί, τους ε, καταβλισμούς τους επισκέφθηκαν και, ε, και πολλοί δωρητές που ήταν, όπου υπήρχε παραδειγματική τάξη και το World Food Program τι να παρέχει φαγητό, έδινε μια κάρτα, φαινόταν σαν πιστοτική κάρτα, έτσι ώστε να πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί στα σούπερ μάρκετ να ψωνίζουν, να νιώθουν ότι εντάσσονται στην καθημερινή ζωή. Επίσης, σε κάθε καταβλισμό υπήρχε μια αγορά όπου ο καθένας μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Είδαμε εξαιρετικά project της UNICEF με παιδιά και ε, πολλά παιδιά τραυματισμένα που έχασαν την οικογένειά τους είδαν ε, φρικαλέα πράγματα, αντίκρισαν φρικαλαιότητες. Ο Σοακίν ε, επισκέφθηκε ε, τις οικογένειες με, μια οικογένεια με παιδιά, τις οικογένειες με παιδιά, εγώ δεν πήγα εκεί, αλλά ε, βρίσκονται εκεί τρία χρόνια και δεν βλέπουν να διαγράφεται καμία ελπίδα να επιστρέψουν στη Συρία. Δεν έχουν άδεια Εργασία στην Τουρκία και το θέμα αυτό απασχολεί την τουρκική κυβέρνηση και είναι ένα σημείο διελκυστίνδας ε, στα πολιτικά κόμματα. Μιλάνε για επισκέπτες. Καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ντόπιου. Υπάρχει κάποια αντιδικία. Η ΤΕΠ έχει ένα 1.400.000 ανθρώπους. Ξέρουμε ότι και εδώ έρχονται πολλοί πρόσφυγες, αλλά δεν βλέπουμε τους αριθμούς που είδαμε στην Τουρκία. Και ο Ενρίκε είπε ότι πώς έχει κατάσταση στο Λίβανο και εκεί είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Έγινε μια πρώτη συζήτηση στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα και μιλήσαμε για τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της ε, προσφυγικής κρίσης. Ήταν πια καιρός για κάτι τέτοιο. Είναι ε, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος γιατί δεν υπάρχει η τάση να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να παραμείνουν στην Ιορδανία, στο Λίβανο, στην Τουρκία. Υπάρχει μία μετακίνηση προς την Ευρώπη, γιατί ένιωσα ότι δεν μπορούν να ενταχθούν εκεί. Αυτό το ζήσαμε και στην Αφρική. Η ύπατη για τους πρόσφυγες το γνωρίζει πολύ καλά αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη χρηματοδότηση. Στην Ευρώπη τα κράτη-μέλη δεν ε, συντονίστηκαν. Ο ένας το, το παρέπεμπε στον άλλον το ζήτημα. Στην Τουρκία είδαμε το, την κορονίδα της αποτυχίας της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και τώρα ε, διπλασιάζεται αυτός ο κόπος σε σχέση με το αν το είχαμε αντιμετωπίσει έγκαιρα το ζήτημα. Αλλά οι φορείς ε, και η κοινωνία των πολιτών συνεργάστηκαν όσο καλύτερα μπορούσαν. Αυτό αφορούσε και τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά πολλά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Gaziantep έστελναν εκθέσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πολλοί που έρχονται σε εμά έρχονται μέσω της ε, Τουρκίας. Έγιναν συναντήσεις με τον Ερντογάν, αλλά όλα αυτά ε, θα έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα. Και βεβαίως και η βομβιστική ενέργεια περιέπλεξε τα πράγματα. Ο Ζακίμ θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν σύντομο το ταξίδι και η αποστολή, αλλά πραγματικά με περιστατικά και εντυπώσει. Και η έκθεση είναι πάρα πολύ λεπτομέρη. μπορείτε να διαβάσετε όλε τι λεπτομέρειε. Θα ήθελα να τονίσω αυτά που είπε η πρόεδρο. Η σύγκρουση στην Συρία, στο Ιράκ δεν είναι κάτι καινούριο. Έχουν ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια και σε ένα βαθμό υποκρινόμαστε ότι αυτό είναι μακριά μας. Στο Φάουστ του Γκέτε αναφέρεται ότι τι με πειράζει και τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο κόσμος στην Τουρκία. Έτσι ήταν και η πολιτική λοιπόν των τελευταίων χρόνων. Μόνο που πλέον στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο η Τουρκία είναι έξω πρωτά μας. Και αυτό βλέπουμε να συμβαίνει τώρα. Η κατάσταση λοιπόν στο νότο της Τουρκίας σαν τα τελικά της Τουρκίας είναι οι εξή. Δύο εκατομμύρια άτομα τα οποία έχουν προσφύγει στην Τουρκία από την Συρία. Δεν μιλάμε για Ιορδανία, Λίβανο. Εκεί υπάρχουν ανάλογα αριθμητικά στοιχεία, αλλά τουλάχιστον ε, περίπου δύο εκατομμύρια στην Τουρκία. 200.000 στα προσφυγικά καταλήμματα. Δεν λέω ότι ζουν εκεί, ενώ ότι είναι κλεισμένοι εκεί, γιατί έχουν τα απολύτως απαραίτητα, αλλά δεν έχουν καμία ελευθερία κινήσεων. Η εκπαίδευση για τα παιδιά, αλλά σήμερα βλέπουμε ότι γίνονται παιδιά στα καταλήμματα αυτά και επαναλαμβάνονται αυτά που πριν από 40-50 χρόνια γίνονται και με τους Παλαιστίνιους στα προσφυγικά καταλήμματα. Αλλά οι πιο πολλοί προτιμούν και έχουν προτιμήσει να μην πάνε στα καταλήμματα αυτά να έχουν μια ελευθερία κινήσεων στις πόλεις, στα χωριά, έξω από τις πόλεις. Όσο η Τουρκία λοιπόν ήταν σε μια κάπως καλύτερη οικονομική κατάσταση, δεν υπήρχαν μεν άδειε εργασίες, αλλά στη μαύρη αγορά απασχολούνταν οι Σύριοι πρόσφυγες και οι άλλοι πρόσφυγες ως φτηνό εργατικό δυναμικό. ήταν μια κατάσταση λίγο πολύ αποδεκτή. Η κατάσταση όμως έχει επιδεινωθεί πλέον στην ε, Τουρκία σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και οι πολιτικές ισορροπίες, όπως είπε και η Πρόεδρος, είναι πολύ ευαίσθητες και ανατρέψιμες. Η αντιπαράθεση λοιπόν μεταξύ του τουρκικού στρατού και των Κούρδων οξύνεται και πάει. Και ασφαλώς ε, η κατάσταση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία περιπλάκεται περαιτέρω. Ναι, μεν ζουν εκεί και εγώ επισκέφτηκα κάποιες οικογένειες και ζουν ε, στο περιθώριο της ε, κοινωνίας, σε γκαράζ, σε γιαπιά και δεν ζουν δωρεάν εκεί, δεν μένουν δωρεάν, πληρώνουν. Νίκια. Νίκια βέβαια θα υπονοήσω ότι υπάρχουν σπίτια. Υπερβολικά μεγάλα ποσά Όποιοι έχουν κάποια υποστήριξη από το εξωτερικό, κάπως τα βγάζουν πέρα. Όποιοι δεν έχουν υποστήριξη τέτοια, για αυτούς τα πράγματα περιπλέκονται πολύ. Και σε αυτού προσθήκονται και τα άτομα τα οποία έχουν συμμετάσχει στον πόλεμο, έχουν πληγωθεί, έχουν τραυματιστεί. Εγώ επισκέφτηκα δύο οικογένειε και είδα ε, ένα νερό κορίτσι με ακροτηριασμένα άκρα έναν πατέρα που δεν είχε καν τα βασικά όταν ε, βρέθηκε ε, σε νάρκες και δεν μπορεί πλέον να εργαστεί. Είναι λοιπόν όλο και πιο οξυμένη η κατάσταση έκ της ανάγκης ε, εκεί. Η υποστήριξη δε την οποία παρήχε ως τώρα η Τουρκία δεν μπορεί να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου στα ίδια επίπεδα. Άρα το ερώτημα που ανακύπτει για αυτά τα άτομα είναι πού θα πάνε. Πήγα μέχρι τα όρια, μέχρι τα σύνορα με τη Συρία. Είναι κλειστά τα σύνορα πλέον, τα έχουν κλείσει οι Τούρκοι. Αν κάποιος έρθει από το Αλέπι, από το Όλμς και έχει διαπιστωθεί βομβιστική ενέργεια και είναι σαφές ότι το άτομο αυτό έχει τραυματιστεί λόγω της βομβιστικής αυτής ε, επίθεσης. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν τους αφήνουν να μπουν. Ιδάλλως κλειστά τα σύνορα. Η πρόεδρος, η Λίντα, είπε ότι για να μπει κανεί ε, σε ένα προσφυγικό κατευλισμό θα πρέπει να καταχωριστεί και να περιμένει εβδομάδες ολόκληρε στο Υπουργείο Ιστορικών. Μου απαγόρευσαν λοιπόν ε, και μένα να έχω πρόσβαση στα καταλήμματα αυτά, στους καταβλισμούς, γιατί, για τους γραφειοκρατικούς αυτούς λόγους. Όσοι ήρθαν από τη Συρία στην Τουρκία, ε, έχουν ένα ιδιαίτερο καθεστώς στην Τουρκία. Το θεωρούν ε, προσκεκλημένους. Έχουν ιδιαίτερο καθεστώς για το Αλέπι, για την Όλυμψη, για την Βόρεια Συρία υπάρχει η αίσθηση ευθύνη, ε, σαν να ήταν τμήμα του, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ακόμα αυτή. Αλλά στο Καζιαντέπ ε, είδαμε και πολλά άτομα από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ, από το Πακιστάν. Αυτούς δεν τους φροντίζουν. Δεν έχουν αυτό το ιδιαίτερο καθεστώ. αυτοί. Οι Ιρακινοί που ήρθαν πριν από δύο-τρία χρόνια δεν τους επιτρέπουν οι δεκινές αρχές να επιστρέψουν, γιατί τους ρωτάνε με τι χαρτιά φύγατε και γιατί να σας δεχτούμε τώρα πάλι πίσω. Και έτσι λοιπόν ε, η κατάσταση είναι περίπλοκη. Για αυτά που βλέπουμε στην ε, Γερμανία, στην ε, Ευρώπη, ο κόσμος χάνει την ελπίδα του, την έχει ήδη χάσει την ελπίδα του να επιστρέψει στην πατρίδα του. Γιατί συνεχίζεται η σύραξη. Και άρα, ε, όσο δυσκολεύει και η επιβίωσή τους στις χώρες υποδοχής, η λύση ποια είναι. Είτε οι νέοι να προσπαθήσουν να βγάλουν χρήματα κάπου αλλού, προκειμένου να θρέψουν αυτούς που έχουν μείνει στην Τουρκία, για παράδειγμα. Και αν δεν φτάνουν τα λεφτά αυτά, αναρωτιέμαι τι θα κάνει ο κόσμος αυτός. Για να μην συζητήσουμε για την ε, ροή προσφύγων που θα συνεχιστεί ασφαλώς. Όσο εκ του πιστεύουμε ότι τέσσερα θέματα θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Το θέμα είναι το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας επιτόπου. Ιδιαίτερος αναφέρθηκε το θέμα της ε, υγειονομικής περίθαλψης. Πάρα πολύ σημαντικό. Τόσο μεγάλη ομάδα ανθρώπων. <coughs> Χρειάζεται υποστήριξη υγεία τους. Το θέμα της νέας γενιάς, η εκπαίδευση. Και ασφαλώς αυτό αφορά και την επιβίωσή τους και την ε, διαποριστική τους δραστηριότητα. Ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Εν τω μεταξύ, πολλά κράτη, όχι μόνο κράτη-μέλη, αλλά όλοι όσοι συμμετέχουν στη σύγκρουση αυτή με οποιαδήποτε μορφή, θα πρέπει σίγουρα να δραστηριοποιηθούν και σε ό,τι αφορά την εξωτερική της πολιτική, προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις. Γιατί είναι προβλέπω ότι μόνο θα αυξηθούν οι δυσκολίες και για μας. Και δεν θέλω καν να σκεφτώ σε αυτή τη φάση ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες. Σας ευχαριστώ. Θέλει κανένα συνάδελφο να κάνει ερωτήσεις, να θέξει κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώχαν, για τα σχόλια αυτά. Χτες παραβρέθηκα στην Γερμανία σε ένα ε, καταβλισμό μεταναστών. Και είναι σε σαφές ότι πολλοί προσπαθούν να ξεφύγουν και από την στρατολόγηση του Ασάντ. Μα είπαν ότι είναι καλή υποστήριξη γενικά, αλλά αυτό που μου είπαν ότι οι πιο πολλοί έχουν οικογένεια όχι στα στρατόπεδα, όχι στους καταβλισμούς, αλλά στη Συρία. Μεγάλη μερίδα λοιπόν, δεν έχω τα επίσημα στοιχεία, ούτε τα στατιστικά στοιχεία, προσπαθούν να φέρουν και τις οικογένειές τους εδώ, να τους φέρουν από τη Συρία. Δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το αριθμό. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Πιο πολλοί έχουν και παιδιά. Αυτοί οι νέοι λοιπόν ως επιτοπλίστων έχουν και οικογένειες. Είναι μεγάλη η ανθρωπιστική λοιπόν κρίση, η οποία θα μπορούσε να προκύψει μόνο και μόνο από αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τη σχετεύσουμε και να βρούμε άλλους τρόπους ανθρωπιστικής βοήθειας. Ακόμα και για άτομα που ζητούν ε, άσυλο ως πρόσφυγες ή πρόεδρος. Ναι, οι πιο πολύ εκτοπισμένοι είναι ιστορικά εκτοπισμένοι στη Συρία. Έγινε γύρω στρογγυλής τραπέζης με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στη Συρία προκειμένου ο κόσμος να ξέρει τι κίνδυνο τρέχει, να ξέρει τι ανθρωπιστική βοήθεια υπάρχει. Είναι τεράστιο λοιπόν το πρόβλημα αυτό. Είναι πραγματικά μεγάλα τα προβλήματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο κύριος Νόιζερ. Ο κύριος η Λίντα και εγώ ε, συζητούσαμε, συζητήσαμε και μιλήσαμε για την κατάσταση των σύρων προσφύγων στην Τουρκία. Αυτό είναι ένα τμήμα μόνο του προβλήματο. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν και πολλοί Ιρακινοί. Και δεν έχουν ε, ησυχάσει τα πράγματα σε καμία περίπτωση στο Ιράκ. Θα έρθουν και άλλοι και από το Αφγανιστάν. Γιατί και εκεί η σύραξη έχει οξυνθεί. Η κατάσταση στο Κούντος, όπου 600 Ταλιμπάν κατάφεραν να διώξουν 7.000 στρατιωτικούς Αφγανούς από την πόλη. Ήμουν λοιπόν στην, Ανατολική, στην Κεντρική Ασία, όπου και ετοιμάζονται η επόμενη κρίση. Εκατομμύρια άνθρωποι από την Κυργιστία από τον Τεδικιστάν, από το Ουσμπεκιστάν βρίσκονταν στην Ρωσία ως ε, φιλοξενούμενοι εργαζόμενοι, γκαστραμπάιτερ, α το πούμε έτσι. Και με το, πτώση του στο ρούβλι, πλέον δεν έχουν χρήματα να στείλουν στους, στις οικογένειές τους. 50% λοιπόν ε, της οικονομίας του Σαντζικιστάν ήταν από εμβάσματα. Αυτό πλέον σταματάει. Τι σημαίνει αυτό με τη σειρά του? Ότι πολλοί από τους νέους αυτούς άνδρες 20 έως 50 ετών τα στραφούν αλλού. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ένα πρόβλημα μεμονωμένο. Όχι. Υπάρχουν πολλοί ομόκεντροι κύκλοι και αυτοί φτάνουν μέχρι και την Ασία, μέχρι και την Αφρική. Σε περίπτωση και περαιτέρω ενδεχόμενων συγκρούσεων. Yeah, thank you. Um... Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλει κάτι να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και την Επιτροπή, την ε, Επιτροπή που παρευρέθηκε στην, ε, Άγκυρα και, στην, ε, και στον Γκάζιεντεπ. Ε, όταν μιλάω για αποτυχία της πολιτικής, ε, δεν μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μιλάω για την Επιτροπή. Η Επιτροπή εκεί γνώριζε πολύ καλά την κατάσταση. Δυστυχώς όμως το Συμβούλιο δεν ε, εισάκουσε την κατάσταση μέχρι ότου έφτασε πρώτον πυλών της. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ. Ε, έχουμε από κάποια Γενική Διεύθυνση Επιτροπής, η Γενική Διεύθυνση ΝΙΕ και θα ήθελα να μου πείτε τι κάνετε ως προς την πολιτική γειτονίας. Ο κύριος ε, Πατρίκ και ο κύριος Καλοσκάνο από τη Γενική Διεύθυνση ΝΙΕ και η Λετίτσια Μοντεκάλβο από την ΕΚΟ. Ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Θέλετε κάτι να πείτε. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιος από την ΕΕΔ εδώ έτσι κι αλλιώς. Εγώ είμαι η κυρία Μοντεκάλβο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεσή σας. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω από πλευράς ε, των συναδέλφων που ασχολούνται και με τις ε, ε, διασυνοριακές ε, μεταφορές από την Τουρκία και ιδιαίτερα στην Καζιαντέπ. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Σύριοι πρόσφυγες στην Τουρκία. Μιλάμε για 500.000 παιδιά που δεν παρακολουθούν σχολείο, δεν έχουν κάποια εκπαίδευση και δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και συνεπώς οι Σύριοι δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για εργασία. Έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς, μαύρη εργασία και ούτω καθεξής. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ είναι το εξής. Οι ανάγκες στην Τουρκία αυξάνονται, αλλά λόγω λιτότητας του προϋπολογισμού δεν μπορούμε να παράσουμε τα πάντα σε όλους. Αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει 36 εκατομμύρια για να υποστηρίξουμε του Σύριους πρόσφυγες ε, στην Τουρκία για το σύστημα υγείας, την αναπαραγωγική υγεία, την εκπαίδευση, διατροφή. Για να βοηθήσουμε τα παιδιά και τους δασκάλους ε, για να έχουν μία ποιοτική εκπαίδευση 7.000 παιδιά, για παράδειγμα, και αυτή τη στιγμή συζητάμε μία, για μία επιχείρηση διάσωσης με την ακτοφυλακή. και επειδή έγινε ε, λόγος για επιπρόσθετα χρήματα για το Ιράκ, δώσαμε χρήματα σε ε, φορείς των Ηνωμένων Εθνών και ΜΚΟ Και για τη διατροφική βοήθεια υπάρχει μια πιλωτική πρωτοβουλία για ειδικά βάουτσερ, για ε, διατροφή, για τροφή μέσα στους ε, καταβλισμούς. Γιατί περισσότεροι βρίσκονται σε ε, αστικό περιβάλλον ή αγροτικό και δεν βρίσκονται μέσα στους καταβλισμούς που διαχειρίζεται η δια Διασυνοριακά μέχρι τώρα για το 2015 το οικονομικό έτος δόθηκαν 70 εκατομμύρια ευρώ για διασυνοριακή βοήθεια και 42 εκατομμύρια στην Τουρκία για ε, ή να υπάρχει πρόσβαση στο Αλέπο, στη Λατάχια, στη Λατάκια και γενικά στη Βόρειο Συρία όπου υπάρχουν ευρύτατες σειράξεις και βεβαίως προστασία και πρόσβαση στην υγεία. Γιατί αν θέλουμε να φτάσουμε στους πιο ε, ευάλωτους θα πρέπει να ξέρουμε ότι 400.000 πρόσφυγες βρίσκονται σε ε, περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τους ευάλωτους, τις ευάλωτες κατηγορίες. Από την Γενική Διεύθυνση Νία, Γειτονία και Διεύρυνση, εγώ προέρχομαι, Κάρλος Κάνο, προέρχομαι από την Γενική Διεύθυνση ΝΙΕΡ. Ο κύριος Πακέ που έπρεπε να ε, είναι εδώ έχει πολλές συναντήσεις λόγω των τραγικών γεγονότων στην Άγκυρα το Σαββατοκύριακο και οποιαδήποτε στιγμή μαζί με τους ε, συναδέλφους ε, θα σας εκθέσουμε την κατάσταση όποτε επιθυμείτε, αλλά σήμερα ήταν αδύνατον. Όποτε όμως το επιθυμείτε μπορούμε να το κάνουμε. Ξέρω ότι και εσείς ασχολείστε με την ανθρωπιστική βοήθεια. Είδαμε πώς διαχειριζόσαστε τα, τα κονδύλια για την πολιτική γειτονίας θα μας απασχολήσει το θέμα δυστυχώς και στο μέλλον και θα δούμε τι θα γίνει με την Τουρκία στο εγγύς μέλλον. Και φτάνουμε στο σημείο 6 που είναι η κατάσταση της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση. Η ε, Μπεθέρα Μπαστερετσέ έχει συντάξει μία έκθεση και επίσης και η ΛΥΜΠΕ για την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη μιας ε, ολιστικής προσέγγισης. Η ΛΥΜΠΕ άλλαξε την προθεσμία, θα ε, ψηφίσουμε το Δεκέμβριο, άρα έχουμε λίγο χρόνο για να συνεργαστούμε με τα μέλη μας και να φτάσουμε σε συμβιβασμούς. σε συνεργασία με τη ΛΥΠΕ. Η κυρία Μπεθέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους φίλους από τις πολιτικές ομάδες γιατί έχουν καταθέσει πάρα πολλές εκατοντάδες τροπολογίες έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για ένα θέμα το οποίο είναι απαραίτητο να συζητήσουμε και το οποίο θα μπορέσει να βελτιωθεί με τη δική του συνεισφορά. Θα επηρεάσουν το περιεχόμενο λοιπόν και το ύφος του κειμένου μέσω των τροπολογιών. Θα παρουσιάσουμε συμβιβαστικές τροπολογίες. Νομίζω ότι ε, η γνωμοδότηση αυτή έχει στενή σχέση με την έκθεση της ΛΥΜΠΕ Ξεκινήσαμε λοιπόν με την απόφαση του Νοεμβρίου ή μάλλον θα έχουμε την προθεσμία του Νοεμβρίου. Η συνάντηση η κοινή αυτή θα είναι πολύ σημαντική για να καταλήξουμε στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Αυτό θα δείχνει το, την κοινή προσπάθεια που κάνουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ανάπτυξης. Είμαι στη διάθεση όλων των συναδέλφων για να συνεχίσουμε να συνεργαστούμε στο κείμενο αυτό και τον μήνα Νοέμβριο ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα έγγραφο ισχυρό, ενδιαφέρον και με συγκεκριμένες προτάσεις για το τι θα πρέπει να κάνουμε γύρω από το πρόβλημα. από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Να ευχαριστήσω επίσης και τους άλλους συναδέλφους που με τη δική τους συνεισφορά κατέθεσαν τις τροπολογίες τις οποίες ε, αναφέρθηκε η ομιλήτρια. Ελπίζω να καταλήξουμε σε έναν ικανοποιητικό αριθμό συμβιβαστικών προτάσεων. Είναι εξής, τα εξής θέματα αυτά τα οποία με ενδιαφέρουν. Ο ορισμός του ε, συγκεκριμένου έφραυστου προσώπου. Δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στα παιδιά και τις γυναίκες, αλλά επίσης και τους ηλικιωμένους και αυτούς οι οποίοι έχουν ειδικά χαρακτηριστικά και ειδικέ ανάγκες. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να τροπολογηθεί είναι η στήριξη της συνεργασίας με τρίτες χώρες, χώρες προέλευσης και χώρες διαμετακόμισης έχει παρουσιαστεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη μετανάστευση. ζητώντας, ε, θέτοντας πλέον ως ανδιαφυσβήτητη ανάγκη την αναθεώρηση ε, του Δουβλίνου 2. Θα πρέπει οι αποφάσεις οι κοινοτικές θα είναι ε, υποχρεωτικές για τα κράτη-μέλη ένα κοινό ευρωπαϊκό επίσης σύστημα για τον τομέα του ασύλου. Είναι ένα θέμα στο οποίο, με το οποίο έχουμε ασχοληθεί ε, πάρα πολλά χρόνια και χωρίς δυστυχώς πολλά αποτελέσματα. Και τέλος θα πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε θα πρέπει να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους πρόσφυγες με αξιοπρέπεια και με σεβασμό στα αναφέρετα δικαιώματά τους και ταυτόχρονα να μιλήσουμε για τον μηχανισμό αναθεώρησης ε, των κανονισμών που ισχύουν για την αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, επόμενος μιλητής, ο κύριος Σαλόμ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να πάρω το λόγο αντικαθιστώντας την Έλλη Σλάιν, η οποία είναι σκιώδηση συγγήτρια της πολιτικής μου ομάδας για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση από κοινού το σύνολο των Ιταλών συναδέλφων. Έχει πάει στη Ρώμη η κυρία Σλάιν ε, και θα γίνει δεκτή από τον ε, πρόεδρο της ε, Ιταλικής Δημοκρατίας. Ελπίζω να πω αυτά τα οποία θα ήθελε και αυτή να πει. Να ευχαριστήσω την Πεατρίση για την συγγραφή της γνωμοδότησής της. Έχουμε ήδη συναντηθεί και έχουμε ανταλλάξει απόψεις έχει μεγάλη σημασία η μεταναστευτική κρίση στην Μεσόγειο. Δεν είναι μια κρίση η οποία άπτεται μόνο των νομικών προοπτικών της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, αλλά επίσης αναφέρεται και σε θέματα αναπτυξιακά και σε θέματα προστασίας των μεταναστών. Από πλευράς της κυρίας Σλάιν θα ήθελα να πω ότι συμφωνεί με την Πεατρίς ότι το θέμα για την, της βοήθειας για την ανάπτυξη περιλαμβάνει την καταπολέμηση των ριζών των προβλημάτων που προκαλούν την μετανάστευση και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει ένα σύνδεσμος υποχρεωτικά ανάμεσα στις αναπτυξιακές πολιτικές από τη μία και τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουμε στο μεταναστευτικό πεδίο από την άλλη δεν θα διαφωνήσουμε ότι οι αιτίες οι οποίες προκαλούν τη μετανάστευση μπορούν να επιληθούν με αναπτυξιακή προοπτική. Αλλά ταυτόχρονα όμως και οι αναπτυξιακές πολιτικές δεν θα πρέπει να δημιουργούν τροχοπέδες στους κατοίκους περιοχών που για διάφορους λόγους θέλουν να μεταναστεύσουν αναζητώντας περισσότερες ευκαιρίες και να βελτιώσουν την ζωή τους. Η ανάπτυξη δηλαδή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κατάσβεση της επιθυμίας της μετανάστευσης εκεί όπου είναι δικαιολογημένη και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο των συνόρων που πολλές φορές συνεπάγεται την αύξηση του κινδύνου για τους πιθανούς μετανάστες. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε στη σταθερότητα των περιοχών τις οποίες ε, ε, θέλουμε να βοηθήσουμε ελέγχοντας ε, τις εξελίξεις έτσι ώστε και τα χρήματα τα οποία δίδουμε να χρησιμοποιούνται σωστά και θα πρέπει να πηγαίνουν απευθείας στα άτομα τα οποία ε, έχουν ανάγκη τα χρήματα αυτά, διότι πάρα πολύ συχνά τα πρόσωπα αυτά είναι θύματα των κυβερνήσεων ε, που είναι υπεύθυνες για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα presentar la ponente eh, en la sombra de mi grupo, algunas de las cuales yo, Enrique Guerrero, también firmo, eh, abordamos la cuestión de las remesas, ε, Ζητάμε λοιπόν να μεγιστοποιήσουμε την βοήθεια για την ανάπτυξη και να προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε επίσης και το κόστος για τις επιστροφές της επαναπροωθήσεις σε βάση περιπτώσει των προσώπων αυτών στις χώρες προέλευσης. Είναι 100 περίπου οι τροπολογίες αυτές. Νομίζω ότι η Μπεατρίς θα τις αντιμετωπίσει με ε, αισιόδοξο τρόπο και στο τέλος ελπίζω ε, θα έχουμε πολύ λιγότερες τροπολογίες όταν καταλήξουμε στην Ολομέλεια για μια γνωμοδότηση η οποία θα είναι θετική γιατί θα δίνει την δυνατότητα να ξεφύγουμε από τα τεχνικά βασανιστήρια των ψηφοφοριών βοηθώντας ε, και την εισηγήτρια, βοηθώντας και τη διεξαγωγή, ε, τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών. Αυτό το οποίο εν πάση περιπτώσει έχει σημασία, λέει ο κύριος Σαλόμ, είναι ότι θα πρέπει να καλύπτεται από την θέση της ΛΥΜΠΕ η οποία λέει ότι για να αντιμετωπίσουμε τη μεταναστευτική κρίση δεν απαιτούνται μόνο διακανονιστικές λύσεις, μεθοριακές ρυθμίσεις, αλλά απαιτείται όμως και προσπάθεια καταπολέμησης των αιτιών που δημιουργούν στις μεταναστευτικές ροές και οι οποίες με τη σειρά τους είναι συνδεδεμένες με τις αναπτυξιακές πολιτικές τις οποίες έχουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Um, Κύριε Σαρτζοντίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και για την εισαγωγή που κάνατε για την ε, επίσκεψη την αποστολή στο Γκαζιαντέπ. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η παρουσίαση των όσων ζήσατε. Ευχαριστώ και τον Ισή για την Πεσέρα. Δεν ξέρω κατά πόσον το είδατε. Ήρθατε αντιμέτωποι με αυτό. Αλλά και ξεχάγεται εδώ και καιρό μία συζήτηση από την Επιτροπή Ανάπτυξης με άλλους φορείς για το κατά πόσο η αναπτυξιακή βοήθεια να χρησιμεύει, είναι χάσιμο χρήματο. Όσοι λένε ότι είναι χάσιμο χρήματο και θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο πολύ το εμπόριο για την αναπτυξιακή βοήθεια είναι σπατάλη χρημάτων μόνο. Αυτοί λοιπόν τώρα λένε ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε να αυξήσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια, γιατί αυτό θα σταματήσει τι μεταναστευτικέ ροέ. Αυτό είναι μύθος, ξέρετε. Κάθε φορά που βελτιώνεται η οικονομία κάπου, αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερε μεταναστευτικέ ροέ. Δεν είναι πρόβλημα αυτό βέβαια, αλλά καταδεικνύει ότι η αύξηση τη οικονομία δεν σταματάει απαραίτητα τι μεταναστευτικέ ροέ, αλλά ίσω και να επιτρέπει στον κόσμο να φύγει από εκεί που είναι. Αυτό που επίσης διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχουν κανόνες για το πόσο δαπανάται η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια από τον ΆΣΑ και την Επιτροπή που μας επιτρέπουν να χρηματοδοτούμε καταλήμματα σε δικέ χώρες από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και αυτό το βλέπω και στη χώρα μου. Είμαστε περήφανοι που Είμαστε στο 0,7% πριν από κάποια χρόνια των ετήσιων δαπανών μας και τώρα μειώθηκε το ποσό αυτό και τώρα πάλι είμαστε στο 0,7% γιατί ξοδεύουμε πιο πολλά χρήματα για την υποδοχή κόσμου και την παροχή καταλήμματος σε ανθρώπους μέσα στις κατοχώρες, στην επικράτειά μας. Μια γνωμοδότηση λοιπόν από την Επιτροπή Ανάπτυξης είναι σημαντική η έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Όχι μόνο για να τονίσουμε ότι υπάρχουν πρόσφυγες πιο ευάλωτοι από άλλους, αλλά λόγω του μεγάλου μακροοικονομικού ζητήματος, του πώς χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε την αναπτυξιακή βοήθεια και μήπως θα υπάρξει κατάχρηση του επιχειρήματος της ε, των μεταναστευτικών ροών και τη διακοπή αυτών. Με αυτή την προσέγγιση λοιπόν εξετάζω το κείμενο. Σε λίγε εβδομάδε έχουμε και τη διάσκεψη στη Βαλέτα, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνδεθεί με εκπροσώπου των χωρών τη Αφρική και εκεί θα δούμε λοιπόν πώ η αναπτυξιακή βοήθεια μπορούμε να δώσουμε στι χώρε αυτέ για να σταματήσουν να στέλνουν μετανάστε. Δεν θα βοηθήσει αυτή η προσέγγιση οι ιδέε που θα πρέπει να συνδυαστούν σε ό,τι αφορά τι συμφωνίε, επανειστοχή με την αναπτυξιακή βοήθεια και αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο δρόμο, Η αρχή του more for more που εφαρμόζουμε για τις χώρες που βελτιώνουν την καλή διακυβέρνηση. Όλοι, σε όλους αρέσει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μετέφρασε το Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα ότι το more for more θα μπορούσε να είναι και λίγο ασφαλέ. δηλαδή ε, λιγότερο για λιγότερο. Δεν θα βοηθήσει την κατάσταση. Άρα, προκειμένου στην Επιτροπή Ανάπτυξη να καταρτήσουμε μία γνωμοδότηση η οποία θα έχει κάποιο αντίκτυπο, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο θέμα τη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Πώ θα χρησιμοποιείται και να διαλύσουμε κάποιου μύθου σε ό,τι αφορά τη μείωση τη μετανάστευση με την αύξηση αναπτυξιακή βοήθεια. Γιατί με τον τρόπο αυτό δεν θα είναι ποτέ βιώσιμη η αναπτυξιακή βοήθεια. Εντάξει να ευχαριστήσω την Μπεατρίθ και εγώ από τη δική μου πλευρά. Ήδη είχα εξηγήσει τη θέση του ΕΛΚ. Θα ήθελα να προσθέσω εντάχει ότι από πλευράς προθεσμίας για τις τροπολογίες μέχρι τη ψηφοφορία θα υπάρχουν και επικαιροποιήσεις τη συναντήσει των σκιωδών. Για παράδειγμα, στο κείμενο βλέπουμε την ατζέντα μετά το 2015 που στο ε, μεταξύ έχει αλλάξει σε ατζέντα μέχρι το 2030. Ε, έγινε λόγος και για το ε, Διαφρικανικό Ταμείο και θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε μια νέα συνένεση για την ανάπτυξη. Ελπίζω να τα δούμε όλα αυτά στη συνάντηση των σκιωδών. Μπορούμε να βρούμε ένα μηχανισμό αν συμβαίνουν, αν έχουμε νέα στοιχεία έτσι ώστε να δώσουμε ε, μία περαιτέρω προθεσμία. Μπορούμε να το κάνουμε δημιουργικά. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κείμενα τα οποία δεν είναι ε, επικαιροποιημένα. Η Επιτροπή. Η Επιτροπή. Η κυρία Σουάρες από την DG Home και από την άλλον έναν συνάδελφο ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Ίσως η Γενική Διεθνήση Home καταρχήν, η κυρία Σοάρης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εντάχει να πω ότι παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εργασίες της ΛΥΠΕΤ καθώς και τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπως και την Επιτροπή Ανάπτυξης φυσικά, για την κατάσταση στη Μεσόγειο. Η άποψή μας είναι ότι χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση, είναι κάτι το απαραίτητο και ήδη το Μάιο 2015 είχε εγκριθεί αυτή η ατζέντα που προβάλλει μία συνολική προσέγγιση για τη μετανάστευση και για τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Θεωρούσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα συνολικό πακέτο με τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές. Βλέπουμε τις ανησυχίες σας και στις τροπολογίες Πολλές τις έλαβε υπόψη η Κομισιόν, θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικές. Το δικαίωμα για άσυλο, για χορήγηση ασύλου ε, έχει εγγραφεί στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θέλουμε λοιπόν να εγγυηθούμε το δικαίωμα για άσυλο. Τα πρώτα hot spots είναι λειτουργικά για να δέχονται τους μετανάστες στα σύνορα και να ταυτοποιούν εκείνους που ε, πρέπει να τύχουν προστασίες ή να επανεγκατασταθούν ή εκείνους που δεν έχουν το δικαίωμα παραμονής στην Ευρώπη. Έχουν αρχίσει οι νέες επανεγκαταστάσεις μετά από τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου και δίνεται προτεραιότητα στους ευάλωτους ανθρώπους. Επίσης, ως προς τις, ε, τα αίτια ή τις ρίζες της ε, μετανάστευσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις αιτίες στις χώρες προέλευσης και ε, διαμετακόμισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βοηθά τον πληθυσμό της Συρίας καθώς και την Τουρκία, ε, Λίβανο και η Ορδανία που βρίσκονται στην ε, μπροστογραμμή. Επίσης θέλουμε να προωθήσουμε μια νέα πολιτική, πολιτικής ε, μετανάστευσης και μέχρι το Μάρτιο του 2016 θα προβάλλουμε ένα νέο νομικό πακέτο με βάση την οδηγία για την ε, μπλε κάρτα για τους επιστήμονες και φοιτητές που τώρα συζητείται σε τριμερείς διαλόγους για να στοχεύσουμε σε αυτές τις σημαντικές ομάδες. Σας ευχαριστώ και βεβαίως προσμένουμε την τελική σας έκθεση. Από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ θα... δεν έχετε κάτι να προσθέσετε. Ωραία. Η κυρία Μπεθέρα. Απλώς να ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία τους και πίστη πιστεύω ότι θα πρέπει στο μέλλον να φτάσουμε σε μία ενδιαφέρουσα έκθεση που να αποτελεί πραγματικά προσθέμενη αξία. Χρειάζεται ενημέρωση των στοιχείων και με τη γραμματεία θα συνεργαστούμε στενά έτσι ώστε το κείμενο να είναι επικαιροποιημένο. Και επιμένω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα καλό κείμενο, ένα συνενετικό κείμενο και πιστεύω ότι την προσεχή συνεδρία θα φτάσουμε σε ένα απτό αποτέλεσμα με τροπολογίες συμβασμού που όπως είπε ο Ενρίκε θα πλουστεύσουν την ψηφοφορία αλλά και θα πολύ πιο ευτυχείς όταν θα ψηφίσουμε τροπολογίες συμβασμού οι οποίες είναι ενισχυμένες. Δεν πρέπει σε κάθε τροπολογία να λέμε τα πάντα. Θα πρέπει να αρκεστούμε στην εντολή μας. Δεν χρειαζόμαστε πολλές αιτιολογικές σκέψεις, γιατί διαφορετικά χάνεται το μήνυμα. Το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, όπου είχαμε πολλές ε, τμηματικές ψηφοφορίες. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε σαφείς για το τι θέλουμε σε συνεργασία με τη ΛΥΜΠΕ. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην επαναλαμβάνουμε αυτά που λέει η ΛΥΜΠΕ και τούμπαλιν. Έτσι ώστε να είναι σαφές το μήνυμα και να βοηθήσουμε τον, την εισηγήτρια, η οποία έχει εστιάσει πολύ σωστά την προσοχή της εκεί που πρέπει. Στις 10 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στο τελευταίο θέμα. Ε, απλώς θα ήθελα να σας πω ότι αύριο στις 9.30 θα συναντηθούμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια και θα συζητήσουμε ή για την εφαρμογή των στόχων για την βιώσιμη ανάπτυξη. Οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη ήταν ένας από τους στόχους μας. Ο κύριος Στίερ θα μας πει πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Uh, thank you, Chair, and... Uh, Ευχαριστώ πάρα. Η Σύνοδος στη Νέα Υόρκη ήταν ε, επιτυχία ήδη από πριν, γιατί το αποτέλεσμα έχει ήδη συμφωνηθεί. Και από αυτή την άποψη δεν υπήρχε άγχος. Γιατί ξέραμε ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για τους 17 βιώσιμους ε, στόχους της χιλιετίας και τους 167 ε, στόχους Έγιναν οι ομιλίε από του αρχηγού κυβερνήσεων και κρατών. Και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι από την άποψη αυτή το, η φωνή του Κοινοβουλίου ακούστηκε και στη Σύνοδο στη Νέα Υόρκη για την Ατζέντα 2030. Ε, το πιο σημαντικό στοιχείο στις συζητήσεις μας ήταν η εφαρμογή και η παρακολούθηση της, ε, των 17 SDGs και το γεγονός ότι είναι καθολική αυτή η ατζέντα και τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη και τα κράτη-μέλη της, αλλά και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ατζέντα. και στη διάρκεια των συναντήσεων μας ε, διαβεβαίωσαν ότι έγιναν σοβαρές δεσμεύσεις για την εφαρμογή της ατζέντα. Είχαμε για παράδειγμα συνάντηση με τον ε, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής Αστρικών ε, Υποθέσεων που μας είπε ότι παρά το γεγονό ότι η καινούργια ατζέντα θα εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου του 2016, γιατί πολλέ χώρε εργάζονταν και εφάρμοσαν τα στοιχεία αυτά στα εσωτερικά του προγράμματο. Ήταν λοιπόν πολύ, συντο... πολύ ωφέλιμες αυτές οι συναντήσεις και η συνάντηση με τον Τζον Πούλενγκερ από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Στατιστική Υπηρεσία, που μιλήσαμε για τους δείκτες, τον οποίο μιλήσαμε για τους δείκτες, για τους επόμενους, ε, τα επόμενα βήματα. Υπάρχουν περίπου 300 δείκτες, μας είπε, αν και ήταν ασφαλώς πολύ επιφυλακτικό γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ακόμα και μέχρι τον Μάρτιο του επόμενου έτους θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα τους δείκτες για την καταμέτρηση των 169 στόχων των 17 SDGs. Αυτά φυσικά θα πρέπει να εγκριθούν και από την έκοση. Το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο συζητήσαμε και σήμερα, και αυτό ήταν προεξέχον ζήτημα στις διμερείς ε, συναντήσεις. Έγιναν διάφορες συναντήσεις με τον Helen Clark της UNDP, με τον αναπληρωτή ε, διευθυντή της Women, με τον πρόσωπο της ε, Διεθνούς Τράπεζας, της Παγκόσμιας Τράπεζας, εκπροσώπου τη ε, Επιτροπή Οικονομικών και Κοινωνικών Ζητημάτων ε, του ΟΗΕ που μας διευκρίνησε πώς θα, κατα... θα παρακολουθήσει ο ΟΗΕ τα ζητήματα αυτά. σε ό,τι αφορά το πολιτικό φόρουμ υψηλού επίπεδου Έγινε και ένα καλό debriefing, θεωρώ, μια καλή ενημέρωση με τον ε, Αντιπρόεδρο Τίμερμαντς και με την κυρία Μοργκερίνη και τον Επιτροπό Μίμητσα στην ε, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συγκεντρώσαμε τα συμπεράσματα όλης της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αντιπρόεδρος Τίμερμαντς νομίζω ότι συμπέρανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δραματίζει ηγετικό ρόλο για την ε, ατζέντα του 2030. Νομίζω ότι αυτά λίγο πολύ συνοψίζουν τις βασικές τους απόψεις. Ε. Τόνισε τη σημασία της συνοχής της πολιτικής και προσωπικά δεσμεύτηκε νομίζω για την αναθεώρηση των ιστορικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένη της νέας ατζέντας 2030. Ο Επιτρόπος Μίμητσα στη συνάντηση αυτή μίλησε για την εκκίνηση μιας διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για μια νέα Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη. Και νομίζω ότι επιπροσθέτως προς αυτά ε, έγιναν και κάποιες συναντήσεις με την ε, Save the Children, Free Sachs. Αναφέρθηκε και η Πέτρη σε αυτά. Με τον ειδικό απεστηλμένο για την μετανάστευση του ΟΗΕ και για την ανάπτυξη με την USAID. με μια ανακυβερνητική οργάνωση Beyond 2015 και νομίζω ότι συνολικά, όπως σας είπα, βασικό στόχος ήταν να δούμε πώς η διεθνή κοινότητα προετοιμάζεται για τη φάση εφαρμογής της πολυφιλόδοξης αυτής της ατζέντας επιστρέψαμε από τη Νέα Υόρκη με μία αίσθηση ότι υπάρχουν ασφαλώς και σοβαρές προκλήσεις αλλά και σοβαρές δεσμεύσεις και ότι σημαντικό κομμάτι της δουλειάς έχει ήδη γίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Κυρίως στη φάση προπαρασκευής των δικτών που θα εγκριθούν από το Μάρτιο και μετά. Ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος Τίμερμαντς είπε ότι θα πρέπει να σπάσουμε και τα σιλό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί τα θέματα είναι καθολικού ενδιαφέροντος και θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία και σε εμά ανάμεσα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Δεν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουν οι πρωθυπουργοί και πρόεδροι που αναλαμβάνουν συνεχώς υποχρεώσεις χωρίς συνέχεια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις προς τον Ταβόρ ή τον προηγούμενο μιλητή. Μπεατρίς, θα ήθελα απλά να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε και η Λίντα. Πρόκειται για πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή της και οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε για να αντιμετωπίσουμε διαφορετικές προοπτικές. Νομίζω ότι τα βασικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει κανείς μετά από τη συνάντηση αυτή και την κορυφή αυτή είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει υποχρεωτικά ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται και δρούν οι κυβερνήσεις. Εμείς έχουμε τα ευρωπαϊκά όργανα, γνωρίζουμε ότι δεν επηρεάζουμε τόσο πολύ ε, τη λήψη των ε, αποφάσεων, αλλά απαιτείται να υπάρχει σωστή και επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει ακριβώς να προσπαθήσουμε να εμπνεύσουμε και να δώσουμε ελπίδες ε, όπως ακριβώς στις συναντήσεις τις οποίες είχαμε με το Save the Children. Νομίζω ότι οι νέοι είναι οι μελλοντικοί ηγέτες και ακριβώς αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ο κύριος Βονβόπ ε, είναι αυτός ο οποίος θα αναφερθεί στο θέμα της ολοκλήρωσης του καταλόγου των δικτών και στον εμπλουτισμό των δικτών στο μέλλον. Έχουν υπογράψει κάποιες συμβιβεστικές προτάσεις στα κράτη, αλλά μιλάμε για μία συνένεση σε επίπεδο διεθνές. Ελείπουν όμως οι τελικοί δείκτες. Για να συμπληρώσουμε τον κατάλογο αυτό, θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης οι κυβερνήσεις. Το θέμα δεν είναι θέμα του αρμόδιου κάθε φορά Υπουργού Ανάπτυξης και Συνεργασίας. Η αηφορία και η ανάπτυξη είναι ένα ενιαίο θέμα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάψιο τρόπο, συνολικό τρόπο από όλες τις κυβερνήσεις. Και θα πρέπει και εμείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όχι μόνο να συνεργαστούμε σωστά, να εμπνεύσουμε και να στηρίξουμε τις κυβερνήσεις μας έτσι ώστε αυτές οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια μας να αναλάβουν τις δικές τους υποχρεώσεις. Περίεργα. Ευχαριστώ. Το πλέον σημαντικό πλέον, τη στιγμή που υπάρχει ε, ένα πλαίσιο στοχοθέτησης, είναι να φτάσουμε στην εφαρμογή βρεθήκαμε στη διάσκεψη στην Αντίσα Μπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης όπου είναι ανάμεικτα τα αποτελέσματα. Υπάρχουν ενθουσιώδη στοιχεία και κινητοποίηση πόρων και από την άλλη πλευρά Μία άλλη πτυχή αφορά την ε, εποπτεία αυτών των αποτελεσμάτων με βάση συγκεκριμένους δείκτες. Θα πρέπει λοιπόν να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι έχει μεγάλη πείρα ως προς την ανάπτυξη και τους σχετικούς δείκτες για την βιώσιμη ανάπτυξη και σε αυτή τη διαδικασία κατάρτισης των δικτών θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να μας πει κάτι το πιο συγκεκριμένο για το πώς σκέφτεται ότι μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την ε, πολυσχηδή εργασία της ε, συγκρότησης, κατάρτισης ε, δικτών ανάπτυξης. Ο κύριος Φοντίνη από την Επιτροπή έχετε κάτι να προσθέσετε. Χωρίς μικρόφωνο, ο μιλητής. Ναι, εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα σε σχέση με, το, με την ίδια τη διάσκεψη ε, κορυφής δεν έχω και πολλά να ακούσω σε σχέση με την ε, συνοπτική εικόνα που μας ε, παρουσιάσατε. πολύ επιτυχής η διάσκεψη. Ήταν μια χρονική στιγμή όπου είχαμε τους περισσότερους αργηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη Νέα Υόρκη και από τον Αύγουστο και μετά ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να έχουμε υποστήριξη της ατζέντα και εφαρμογή της. Αυτά είναι τα μηνύματα που πέρασαν, ιδιαίτερα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς, από την ύπατη εκπρόσωπο, ε, την ε, κυρία Μογκερίνη από τον Επίτροπο Μίμητσα και από τη δική σας αντιπροσωπεία που παραβρέθηκε στη Νέα Υόρκη. Ως προς το ερώτημα που θέσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα καταρχήν να πω ότι φυσικά η εφαρμογή αυτής της ατζέντα είναι πολύ σημαντική και ο ορισμός των δικτών είναι ύψης της σημασίας, διότι αυτό αυτά που μετρώνται πρέπει και να εφαρμοστούν. Όταν διαπραγματευτήκαμε αυτή την ατζέντα στη Νέα Υόρκη είχαμε σαφή στοχοθέτηση αλλά για τους δείκτες αποφασίστηκε να αφήσουμε τον ορισμό τους σε μια διακυβερνητική διαδικασία ε, υπό την αιγίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών. Ε, μέσα στα πλαίσια μιας ε, interagency στατιστικολόγων. Τότε θεωρήσαμε ότι δεν ήταν ε, αποδοτικό να συζητάμε πληθώρα δικτών σε διακυβερνητικό επίπεδο και θα ήταν καλύτερα αυτή η εργασία να επιτελεστεί μέσα στα πλαίσια στατιστικολόγων από όλο τον κόσμο σε τεχνικό επίπεδο. Και στη συνέχεια θα αναπαινθεί το ζήτημα στα Ηνωμένα Έθνη το Μάρτιο και θα συζητηθεί από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία και μέσω της Eurostat και των διαφόρων στατιστικών υπηρεσιών κρατών μελών, 5 ε, ή 6 εξ αυτών που είναι μέλη της Interagency. Η τεχνική αυτή εργασία έχει και μία ε, διάσταση κατάρτισης πολιτικής γιατί θα πρέπει οι δείκτες να εκπροσωπούν το επίπεδο πλούτου. Θα πρέπει να έχουμε συνεπή στάση και την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες οργανώσαμε μία τεχνική συνάντηση των εμπειρογνωμόνων, των κρατών μελών και από πλευράς κατάρτισης πολιτικών και στατιστικής και Eurostat για να ακούσει Eurostat όλες τις ε, πλευρές έτσι ώστε να εκπροσωπηθεί η ευρωπαϊκή θέση. Έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι έχει η διαδικασία. Επιπροσθέτως θα πρέπει να πω ότι όταν μιλάμε για αυτή τη διαδικασία μιλάμε για διεθνώς ε, συμφωνημένους δείκτες. Θα έχουμε και περιφερειακούς δείκτες στη συνέχεια που κάθε χώρα θα καταρτήσει και τους δικούς της, τους εθνικούς δείκτες. Άρα υπάρχουν τρία επίπεδα. Υπάρχουν ε, τρεις ομόκεντροι κύκλοι, ε, περιφερειακοί, εθνικοί και διεθνείς δείκτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Το θέμα με τους δείκτες ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή. Αυτή η δείκτες που είναι υπό ανάπτυξη δημοκρατική λογοδοσία, για παράδειγμα, στα πλαίσια της κυβέρνησης. Αυτά δεν είναι απαραίτητα μετρήσιμα ζητήματα για όλους μας. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Στήρ και πάλι. Αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη που έκανε εξαιρετική δουλειά εκπροσώπηση στην Επιτροπή μα και τον Κρίστη Μαζέρα από το άλλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πραγματικά ε, διοργάνωσε εξαιρετικά το πρόγραμμα. Έχετε και πάλι το λόγο λοιπόν. Ναι, θα πρέπει να συμφωνήσω και εγώ. Να ευχαριστήσω και τον ε, Επιτροπή και τον Κριστιαν για το θέμα των δικτών. Να προσθέσω το εξή. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Στατιστικών Στοιχείων ανεπίσημα εξέφρασε Κάτι που είπε και προηγουμένως ο Ότι προφανώς, ε, παρά το γεγονός ότι υπάρχει τεχνική δουλειά που θα πρέπει να γίνει, υπάρχει και πολιτική εξέταση του θέματος. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε λοιπόν και αυτό νομίζω ανεπίσημα το συζητήσαμε ε, η GN να καταλήξει τελικά σε έγκριση των δικτών από τη Γενική Συνέλευση και η ΕΚΟΣΟΚ φυσικά θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει, αλλά θα πρέπει να το παρακολουθούμε και αυτό. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να προσθέσω. Κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι η στιγμή να το συζητήσουμε, αλλά θα μας περιμένει. Στο μέλλον θα το συζητήσουμε και στους δανειστές. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της διαδικασίας αυτής, την εποπτεία της διαδικασία αυτή. Λίντα. Μιλήσατε για την οργάνωση και του έργου του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει αυτά να ληφθούν υπόψη όταν θα καταθέσουμε την πρότασή μας για το ποιος θα είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής των SDGs. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ήταν πολύ καλή η αποστολή και τώρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Μάλιστα, μια πολύ σημαντική ανακοίνωση για αύριο το πρωί. Ξέρω ότι γίνεται διαβούλευση μεταξύ των ομάδων ή ψηφοφορία αύριο. για την εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου του 2010 σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα θα αναβληθεί. Δεν θα ψηφίσουμε στις 9 λοιπόν αύριο θα ξεκινήσουμε στις 9.30. Κανονικά, με την κοινωνιστική συνεδρίαση για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και τους στόχους βιώσιμης αναπτύξης. 9.30 λοιπόν θα ξεκινήσουμε. Θα λάβατε email. Οι βοηθοί παρακαλώ να ειδοποιήσουν τους βουλευτές τους. Δεν έχουμε ψηφοφορία αύριο το πρωί στις 9. Σημαντικότητα αυτό. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τις σημερινές μας εργασίες και μπορούμε να διακόψουμε. Θα λέμε αύριο στις 9.30 το πρωί. Σας ευχαριστώ. γενικά η Πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς εμείς σας ευχαριστούμε.